Καλημέρα, θα έλεγα να ξεκινήσουμε. Εκτάκτος, έχουμε συνεδρίαση της, ε, συνεδρι... της Επιτροπής μας που κρατά μόνο μισή μέρα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ αποτελεσματικοί στη χρήση του χρόνου. Θα εργαστούμε αναγκαστικά σε αυτή την αίθουσα που συνήθω διατίθεται για διαθεσμικέ ε, συνεδριάσει ή τριλόγου. Τριμερεί διαλόγου, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχετε λάβει το σχέδιο ημερήσια διάταξη και σα ανακοινώνω ευθύ αμέσω ότι με την συμφωνία του εισηγητού που θα είναι μαζί μας σε λίγο, του κυρίου Μπέγκε, τα σημεία 9 και 10 αναβάλλονται. Είναι το περίφημο πακέτο της Λισαβόνας για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα μπορούμε να το συζητήσουμε εύστοχα όταν θα έχουμε τι τελευταίε λεπτομέρειε και από την νομική μα υπηρεσία που ήδη μελετά το θέμα, ήδη έχει δώσει απάντηση στη γνωμοδότηση που είχε ζητήσει ο Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου και η διάσκεψη των προέδρων. Υπάρχουν επιπλέον ε, διευκρινήσει που έχουν ζητηθεί από την Επιτροπή μα, ε, έχει εξεταστεί το θέμα και είναι μαζί μα εκπρόσωποι τη νομική υπηρεσία. Εργάζονται πολύ αποτελεσματικά. Του χαιρετώ, του εύχομαι καλημέρα και θα το συζητήσουμε αργότερα. Για τα υπόλοιπα σημεία τη ημερήσια διάταξη, θα τα εξετάσουμε όπω προβλέπετε. Ίσως όχι ακριβώ τη σειρά που αναφέρονται στο έγγραφο, διότι για λόγους είτε της, του προσωπικού προγράμματο κάποιων εισηγητών, είτε και, και των προσκεκλημένων μας για τη συζήτηση ορισμένων θεμάτων, εκεί θα γίνουν κάποιες προσαρμογές στο πρόγραμμά μας. Τώρα, για τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Έχουν άμεση σχέση, εν μέρη, με την ημερήσια διάταξη. Από τη μια, οι συντονιστές των ομάδων που συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, απεφάσισαν να ξαναδούν το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας του προπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 2012, δεδομένου του χρονοδιαγράμματος που ε, υιοθέτησε το Προεδρείο σε ό,τι το φορά. Ο κύριος Φίλερ θα είναι μαζί μας σε λίγο ούτω ή Το Προεδρείο λοιπόν προβλέπει να υιοθετήσει το σχέδιο εκτιμήσεων τη Δευτέρα 7 Μαρτίου, τα draft estimates. Έτσι λοιπόν οι συντονιστές αποφάσισαν να προτείνουν στο Γενική Γραμματέα, στη Γενική Γραμματεία μάλλον, να παρουσιάσει τι ε, προτάσει εκτιμήσεων αυτέ, το σχέδιο εκτιμήσεων, κατά κατά την επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών στις 9 Μαρτίου στο Στρασβούργο. Και εκεί θα γίνει μια πρώτη συζήτηση για το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Φερνάντες, πάντοτε με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προπολογισμών δηλαδή, 15 και 16 Μαρτίου. Αυτό θα μας επιτρέψει να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια συγγνώμη, την ψηφοφορία σε επιτροπή, σε έκτακτη συνεδρίαση τη Επιτροπή Προπολογισμού στι 24 Μαρτίου το απόγευμα ενώ η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ορίζεται για τις 17 Μαρτίου. Αυτό θα μας επιτρέψει να ψηφίσουμε την έκθεση στην Ολομέλεια του Απριλίου. Εγκαίρος δηλαδή. Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να λάβει υπόψη την δική μας την ψηφοφορία κατά την ε, επεξεργασία του σχεδίου προπολογισμού του 2012 σχέδιο προπολογισμού που θυμίζω ότι είναι ενιαίο πλέον για όλα τα θεσμικά όργανα ε, και κατά αυτόν τον τρόπο υποβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται τι δικέ μα εκτιμήσει, αυτέ που θα έχουμε εγκρίνει με ψηφοφορία. Σε ό,τι αφορά τώρα άλλε ανακοινώσει, σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστούμε σήμερα, ο κύριος Άλβαρο, που είναι σκεώδης συγκεκριτής, για τους φιλελευθέρους θα είναι μαζί μας στις 11 μόλις. Οπότε σας προτείνω να αναβάλουμε την ψηφοφορία για τις ε, κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου έκθεση του κυρίου Φερνάντες να την αναβάλουμε για τις 11. Κοιτάζω και την ε, Φραντσέσκα, ο κύριος Φερνάντες ε, συμφωνούν. Χωζέ Μανουέλ θέλει το λόγο για το σημείο αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω την εξή πληροφορία. Το Προεδρείο την Δευτέρα στις 7 Μαρτίου δεν θα εγκρίνει τις εκτιμήσεις, το σχέδιο εκτιμήσεων. Θα αναθέσει όμως εντολή για τις εκτιμήσεις αυτές. Δηλαδή δεν θα ψηφίσουν πριν την έγκριση των κατευθυντηρίων γραμμών στην Ολομέλεια, όπως θα θέλαμε. Είναι μια μικρή διευκρίνηση. Ενδεικτικά σας το λέω και πληροφοριακά. Θα ήθελα να θυμίσω σε όλους τι εξέφρασαν ως επιθυμία οι συντονιστές στην τελευταία συνάντησή τους ως προς την ανάγκη να επικεντρώσουμε μάλλον να φροντίσουμε να ψηφίσουμε στο δυνατόν νωρίτερα και να ενημερώσουμε να ορίσουμε στο δυνατόν νωρίτερα την ε, στιγμή που θα γίνει η ψηφοφορία και να ενημερώσουμε γέρος τους ε, συντονιστές. Δεν είναι εύκολο για τους συντονιστές να καταφέρουν να είναι παρόντες όλοι όσοι πρέπει να ψηφίσουν εάν δεν είναι γνωστή η ώρα που θα γίνει η ψηφοφορία. Σας ζητώ λοιπόν εκ μέρους όλων να γνωστοποιηθεί εν αυτό το χρόνο. Ε, ευχαριστούμε, Σαλπαντόρ. Νομίζω την επιθυμία σου αυτή τη συμμερίζονται όχι μόνο οι συντονιστέ, αλλά όλοι οι συνάδελφοι εδώ. Έχουμε εξαιρετικά μισή μέρα στη διάθεσή μας σήμερα. Συνήθως όταν γίνεται αυτό ε, η ψηφοφορία γίνεται στο δεύτερο μέρος της ε, συνεδρίασης. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Αντί για τις 9 θα ψηφίσουμε στις 11. Ανάλογα με το τι ζήτησαν και οι συντονιστές. Καθώς και οι συγκητέ και οι σκιώδεις συγκητέ. Όμως η ιδεολογική τοποθέτηση του Σαλβαντόρ είναι προφανώς σημαντική. Συνεχίζω λοιπόν με τις διάφορες τροποποίησεις. Μα ζητήθηκε το σημείο της κυρίας Γιάννης να πριν τις 11 και πριν τις 11 θα δούμε και το σημείο που έχει να κάνει με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης για να υποφεληθούμε της παρουσίας του διευθυντή, ενός από τους διευθυντές. Θυμίζω ότι ο αντιπρόεδρος, αντιπρόεδρος Μαρτίνες Μαρτίνες και ο κύριος Πέτερη θα έρθουν στις 10.30. Θα παρουσιάσουν την ε, έκθεσή τους για τη χρηματοδότηση του σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Εδώ υπάρχει ένα σχέδιο χρηματοδότηση για να καλυφθούν ορισμένε από τι προπαρασκευαστικέ δαπάνε αυτού του σχεδίου. Κάποιε ομάδε έχουν ερωτήσει να θέσουν και μα γνωστοποίησαν ότι θέλουν η ψηφοφορία για αυτή τη χρηματοδότηση να αναβληθεί έω ότου απαντηθούν οι ερωτήσει αυτέ. Θα υποφεληθούμε λοιπόν τη παρουσία ε, του κυρίου Μαρτίνε Μαρτίνε και του κυρίου Πέτεριν για να θέσουμε τι ερωτήσει αυτέ. Θα ήθελα τέλο να επισημάνω ότι σε ό,τι αφορά την εντολή για την δράση τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θυμάστε ότι στη συνεδρίασή μα στι 27 Ιανουαρίου είχαμε εγκρίνει με ευρία πλειοψηφία έκθεση για την εντολή αυτή. Βάσει της απόφασης αυτής και με κάποιες προσαρμογές οι οποίες χρειάστηκαν λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στο, στην νότια πλευρά της Μεσογείου. Η Ολομέλεια ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση την θέση του Κοινοβουλίου. Στις 17 Φεβρουαρίου συγκεκριμένα. Η θέση αυτή είναι πλέον η νέα διαπραγματευτική εντολή του Κοινοβουλίου του οποίου η αντιπροσωπεία αποτελείται από τον εισηγητή και τους όδες εισηγητές. Μόλις είναι δυνατόν, Και επειδή ήδη γίνονται διερευνητικέ συζητήσει, έχουν ε, ξεκινήσει στις 28 Φεβρουαρίου και συνεχίζονται, αυτή η διαπραγματευτική ομάδα θα ξεκινήσει τον επίσημο τριμερή διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα στο ανάλογο επίπεδο για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις της δεύτερης ανάγνωσης. Ο, η μορφή που θα πάρει ο τριμερής διάλογος θα λάβει υπόψη και θα σεβαστεί τις διατάξεις της ε, κοινή συμφωνίας ε, σε ό,τι ορίζει το άρθρο 70 για τους πρακτικούς κανόνες ακριβώς ε, και την εξέλιξη της διαδικασίας με τον σχετικό κανονισμό. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις και σχόλια, να θυμίσω ότι είμαστε στο, σε web streaming σήμερα και έχετε και τις κλασικές ενημερώσεις για την εκτέλεση του προπολογισμού 2010 σε αυτή τη φάση της χρονιάς. Ως προς τα πρακτικά Τις προηγούμενες συνεδρίες στις 26 και 27 Ιανουαρίου, σημείο 3, εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρούνται εγκεκριμένε ως το τέλος της συνεδρίας. Περνάμε απευθείας λοιπόν στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, προετοιμασία του προπολογισμού του 2012. Δίνω αμέσως το λόγο στη Φραντζέσκα Μπαλτζάνη, την εισηγήτριά μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είχα προαναγγείλει στην τελευταία μα συνεδρίαση, στην πρόταση ψηφίσματο που σας παρουσιάζω σήμερα και ελπίζω ότι έχετε χρόνο να μελετήσετε, έχω προσπαθήσει να εντοπίσω και να δώσω έμφαση με περισσότερη σαφήνεια σε κάποια στοιχεία που θα μπορούσαμε ε, να παρουσιάσουμε ως πρώτες μας προτεραιότητες στο πλαίσιο της στρατηγικής για το 2020. Η στρατηγική για το 2020, βάσει της πρότασή μου, είναι η καρδιά της ε, σχέσεις που θέλουμε να εγκαθιδρύσουμε ως κοινοβούλιο ε, σε σχέση με τους εθνικούς προϋπολογισμούς είναι μια στρατηγική ευρύτατη και αρκετά περίπλοκη. Όμω νομίζω ότι αυτό ο πυρήνα τη είναι πολύ συγκεκριμένο και έχει και ιδιαίτερη σημασία σε μια τέτοια χρονική στιγμή. Νομίζω ότι εκεί απαιτείται το περισσότερο έργο και μάλιστα έργο ποιότητα στην Ευρώπη. Περισσότερη δουλειά μάλιστα και σε μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση. Περισσότερη απασχόληση χάρη σε περισσότερε επενδύσει. Οι δύο αυτοί αυτές ε, λέξει κλειδιά, περισσότερη δουλειά και απασχόληση και περισσότερε επενδύσει στην Ευρώπη, θα πρέπει να βρεθούν ε, ω πρώτη μέρημνα στην καρδιά του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να ζητήσουμε και την προστιθέμενη αξία του προπολογισμού αυτού. Αυτό θα είναι και ο καρπό των εντατικών μα προσπαθειών. Η έκθεση λοιπόν αυτή δίνει μεγάλη σημασία στις δύο λέξεις κλειδιά αυτές. Ε, την εργασία και ε, την, ε, τις επενδύσεις που θα πρέπει να βρίσκονται στην καρδιά και των εθνικών προπολογισμών. Οι επενδύσει είναι θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο σε αυτές τις ε, στιγμές κρίσης και λιτότητας, διότι οι επενδύσεις απαιτούν μεγάλες δημοσιονομικές προσπάθειες. Δύσκολο να εξοικονομηθούν τέτοιε προσπάθειες σε στιγμές κρίση. Όμω θα είναι και το μόνο μέσο για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την κρίση και να ανακάμψουμε. Εκεί θα αναζητήσουμε το έδαφο για να διαμορφώσουμε σχέσει συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκού προπολογισμού και εθνικών προπολογισμών. Αυτή θα είναι η πιο χρήσιμη σχέση συνεργασία που μπορούμε να διαμορφώσουμε. Έτσι, στο σχέδιο προπολογισμού το 2012 θα πρέπει να κάνουμε ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Και προ μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Να έχουμε ένα προπολογισμό που να στοχεύει πάνω απ' όλα να δημιουργήσει βιώσιμε στρατηγικέ μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Δηλαδή στατηγικέ, όχι κοντόφθαλμε. Θα πρέπει να ξεκινούμε μέσα από τα δύο κεντρικά θέματα αυτά. Στα πλαίσια τη στρατηγική για το 2020, που ήδη υπήρξε αντικείμενο και άλλη σημαντική ψηφοφορία στην τελευταία ολομέλεια του Στρασβούργου, σε μια απόφαση του Κοινοβουλίου που για άλλη μια φορά επισημάναμε τα μεγάλα ε, θέματα που μα ενδιαφέρουν και το πόσο πλούσια μπορεί να αυτή η στρατηγική, μετά λοιπόν από αυτή την απόφαση θέλαμε ε, αποφάσεις ε, με δυνατότητες ευελιξίας Νομίζω ότι όλοι συγκλίνουμε προ αυτόν τον στόχο να έχουμε περισσότερε επενδύσει και περισσότερη εργασία. Ιδίω στη στρατηγική τη νέα μα βιομηχανική πολιτική. Θέλουμε περισσότερε δεξιότητε στον χώρο τη εργασία και για την νεολαία, διότι αυτό ε, μα απασχολεί πολύ το θέμα τη ε, ανεργία των νέων. Εδώ λοιπόν χρειάζονται πρωτοβουλίε ζωτική σημασία στη στρατηγική του 2020 ε, που καλύτερα από άλλε θα μπορούν να εκφράσουν τη μεγάλη μα στήριξη προ την εργασία και την εργασία καλύτερη ποιότητα θα είναι αυτό ένα θεμελιώδε μέσο για την καλύτερη κοινωνική ένταξη, για να δώσουμε σώμα στις αρχέ αλληλεγγύη που τόσο έντονα διατυμπανίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια τη ίδια απόφαση τίθεται και ένα άλλο θέμα που το θεωρώ και πάλι ιδιαίτερα σημαντικό σε σχέση με τον προπολογισμό μα. και ιδίω για το 2012, γιατί οδεύουμε προ το τέλο του, του τη περίοδου προγραμματισμού του προπολογισμού είναι ένα θέμα σημαντικό, είναι το θέμα της ευελιξίας. Πιστεύω ότι το 2012 ε, προτελευταίο χρόνο και έκτο από τα 7 χρόνια της περίοδου προγραμματισμού θα πρέπει με τρόπο πιο πραγματιστικό να χρησιμοποιήσουμε την ευελιξία και ιδίω την ευελιξία του 5% που μας επιτρέπει το άρθρο 37 της Διαθεσμικής Συμφωνίας. Σήμερα, προς το τέλος της περίοδου προγραμματισμού, θα πρέπει πραγματικά να αναλάβουμε την ευθύνη να χρησιμοποιήσουμε πλήρω τη δυνατότητα αυτή. Όμω υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί ευελιξία που μα επιτρέπονται από τη διαθεσμική συμφωνία. Για την επόμενη περίοδο πραγματισμού γίνονται εργαλεία που από μια συγκεκριμένη σκοπιά Νομίζω ότι έχουμε το καθήκον πλέον να τα χρησιμοποιούμε. Η ευελιξία μέσω των διαφόρων κεφαλαίων είναι ε, δυνατότητε ευελιξία. Διότι τον πρώτο τελευταίο χρόνο του προγραμματισμού, του πολιτού πλαισίου, νομίζω ότι πρέπει με τα μέσα που έχουμε στα χέρια μα να δούμε τι λειτουργήσε και τι δεν λειτουργήσε επαρκώ ε, στην περίοδο αυτή. Θα πρέπει λοιπόν έτσι πιο αποτελεσματικά να επαναπρογραμματίσουμε τις δράσεις μας. Έπειτα υπάρχει και άλλο ένα θέμα που ευρέως έχουμε συζητήσει στην τελευταία μας συνεδρίαση, αυτό των αρνητικών προτεραιοτήτων. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να παραμείνει επιτάπητο ως θέμα συζήτηση. Επιπλέον έχουν ξεκινήσει συναντήσεις με τις αρμόδιες επιτροπές ώστε να ε, δούμε ποιε είναι οι δικέ του μέρημνε ω προ τι τομεακέ προτεραιότητε. Παρόλα αυτά, θέλουμε να ανταλλάξουμε μαζί του και απόψει, ώστε να διαμορφώσουμε ένα πνεύμα προπολογισμού εδώ που να κάνει τον προπολογισμό χρήσιμο και εύστοχο για την στρατηγική του 2020. Για μια Ευρώπη με περισσότερη εργασία και με εργαζομένου και εργασία καλύτερη ποιότητα. Ευχαριστώ. Merci. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κυρία Συγγέντρια και σας ευχαριστούμε για αυτό το ευσύνοπτο ε, και τόσο πλήρες έγγραφο το οποίο συντάξατε. Ευχαριστώ Πρόεδρε που με ξαναβαφτίσατε. Δεν με λένε Τζόρτζο αλλά Τζοβάνι. Τέλος πάντων δεν είναι πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον συνάδελφο Μπαλτζάνη για την αξιέπαινη προσπάθεια που κατέβαλε και την εντατική της ε, μέρημνα να προβλέψει για τον προπολογισμό της ερχόμενης χρονιάς, το 2012, το πλαίσιο της στρατηγικής του 2012. Πλαίσιο για μια στρατηγική διαδικασία που ήδη έχει γκρίνει αυτό το Κοινοβούλιο. Εδώ προφανώς πρέπει να δούμε τι προκύπτει από αυτές τις αποφάσεις. Πώς στρατηγικώς θα ευθυγραμμίσουμε τον ετήσιο προπολογισμό με τις βασικές προτεραιότητες που έχει θέσει το Κοινοβούλιο και η Ευρώπη. Εδώ οφείλω να πω ότι εφόσον αυτό το έγγραφο θα το ψηφίσουμε και στην Ολομέλεια και θα αποτελέσει την ε, βασική ένδειξη για να καθορίσουμε προτεραιότητες ως Κοινοβούλιο για την ερχόμενη περίοδο προγραμματισμού και για τι αποφάσει που θα λάβει σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια επιπλέον προσπάθεια ναι. για να δώσουμε πιο συγκεκριμένε ενδείξει προ την Ευρωπαϊκή ακριβώ αυτή Επιτροπή. Για να δούμε ποιε είναι οι προτεραιότητέ μα. Ακριβώ ε, τα στοιχεία φλέξη που σχετίζονται με τη στρατηγική του 2020 ω προτεραιότητε είναι στοιχεία που θέλουμε να προωθήσουμε. Όμω αυτό το πλαίσιο θα ορίσει νομίζω ένα προπολογισμό που όπω πολλοί θύμισαν θα είναι από πολλέ απόψει ε, προπολογισμό λιτότητα. Θα πρέπει λοιπόν να συγκεντρώσουμε εδώ του ε, πόρου. Είναι δύσκολο να σκεφτούμε και να διαδούμε πώς θα έχουμε ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλειών ως ε, προτεραιοτήτων, ενώ έχουμε έναν τόσο αυστηρό προπολογισμό, περιορισμένους πόρους. Κατά τα άλλα, βλέπω πολύ ευνοϊκά τη μέθοδο που προτείνεται να συμμετέχουν ενεργά οι ειδικευμένε αρμόδιε επιτροπέ. Διότι και με αυστηρό προπολογισμό μπορούν παρόλα αυτά να εξοικονομηθούν πόροι και να οριστούν προτεραιότητε απαραίτητε και χρήσιμε για να μπορέσουμε να επωφεληθούμε αποτελεσματικώ από, από του λίγου πόρου, τα λίγα κονδύλια που ενδεχομένω διαθέτουμε. Όταν, αυξάνονται, όταν μειώνονται μάλλον οι πόροι, πρέπει να τι χρησιμοποιούμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το να συμμετέχουν ω το δυνατόν πιο αποτελεσματικά μπορούν οι αρμόδιε επιτροπέ, νομίζω ότι μπορεί να είναι μια καλή συνεισφορά ώστε αυτοί οι πόροι που διαθέτουμε να χρησιμοποιούνται σωστά. Ευχαριστώ λοιπόν ξανά και για κάποιες συγκεκριμένε αναφορές που γίνονται στην οικονομική διακυβέρνηση, την governance, στον πρώτο χρόνο που ε, κατευθυνόμαστε προς αυτήν την ε, φόρμουλα ευθυγραμμισμού με τους εθνικούς προπολογισμού, θα πρέπει στην Ευρώπη να φροντίσουμε να ελέγχουμε και αυτά τα στοιχεία. Αν και η διάρθρωση του ευρωπαϊκού προπολογισμού σήμερα ίσως δεν είναι καταλληλότερη προκειμένου το σύστημα αυτό να είναι ένα σύστημα που να δίνει μόνο καλά αποτελέσματα και να είναι και αποδοτικό. Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε εντατικά και τους ερχόμενους μήνες. Ευχαριστώ. Merci, cher Ευχαριστούμε, Λεπρόεδρος. Οπότε, μετά από αυτή την διπλή ε, εισήγηση που προέρχεται από την ε, Ιταλία, τώρα θα ανέβουμε λίγο, θα πάμε προς τον ε, Βόρα. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ για να ευχαριστήσουμε για την κυρία Μπαλτζάνη για την τόσο άρτια έκθεση. Ε, έχουν κάποιε παρατηρήσει για το θέμα μα ε, εν γέννη. Νομίζω πάντω ότι καλύπτονται εύστοχα τα ε, σωστά ζητήματα και είμαστε ιδιαίτερω ικανοποιημένοι ότι η στρατηγία το 2020 ε, ε θα, θα, θα καλυφθεί από τον προπολογισμό κατόπιν συζητήσεων και προβληματισμών. Η αλήθεια είναι ότι για την τρέχουσα χρήση έχουμε τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν θα αρκέσει και για το χρόνο και για το 2013. Άρα μπροστά μας έχουμε πολλή δουλειά για να δούμε τι θα κάνουμε. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τις ε, υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει όσον αφορά την συνθήκη της Λισαβόνας. Και έχουμε επικεντρώσει την προσοχή μας στο ότι υπάρχουν κάποιοι πόρε. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα τους κατανείμουμε εκ του νέου με το πολυετές πλαίσιο, μια που είναι δύσκολη δουλειά αυτή. Όμως θα πρέπει να έχουμε ισχυρά επιχειρήματα σε σχέση με τις δυνατότητες ανακατανομής των κονδυλίων. Κάτι άλλο τώρα. Κοιτάξτε, τουλάχιστον στην αγγλική κατοχή του κειμένου, νομίζω ότι η διατύπωση είναι ίσως πιο επιθετική από όσο χρειάζεται. Ίσως θα πρέπει να είναι πιο ήπιος και επικοδομητικός ο τόνος. Άρα να ξαναχτενίσουμε το κείμενο για να δούμε τη διατύπωση για να αποφύγουμε αυτό που είναι πριν τα Χριστούγεννα. Άλλωστε, όπως είπατε, από τον βορρά που προερχόμαστε δεν θα ήταν τόσο αποδεκτός ένας τέτοιος τόνος στη διατύπωση. Έχετε δίκιο. Φυσικά και χρειάζονται περισσότερα χρήματα για την θετική 2020, όμως ε, δεν θα πρέπει να απευθυνόμαστε με αυτόν τον τρόπο και να εξωθούμε έτσι το Συμβούλιο. Τώρα, όσον αφορά το προσωπικό. δεν we should Λέτε εδώ πέρα θα πρέπει να αποφύγουμε τις αυξήσεις προσωπικού. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει αρκετό προσωπικό όσον αφορά την ενώση. Αλλά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον για να μπορέσουμε να ανακατενύουμε το προσωπικό. Συμφωνούμε με τις αρχές αλλά ποτέ δεν καταφέρουμε να, ε, να έχουμε ικανοποιητική ανακατανομή του προσωπικού. Πολύ καλή έκθεση. Και εμείς ίσως υποβάλλουμε κάποιες επικοδομητικές ε, τροπολογίες, τόσο ώστε να μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις προκλήσεις που σας επεσήμανα. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε, λέει ο πρόεδρος, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχετε κάποιες τροπολογίες και έτσι θα μπορούσατε να κάνετε πιο ήπια τη διατύπωση. Το θέμα είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο καθένα ε, αλλιώ εκφράζεται. Ε, δηλαδή, για να σε πάρει στα σοβαρά, σε μερικές χώρε πρέπει να τα πει σωμά. Όχι, όχι, δεν λέω ότι αυτό έκανε η Φραντζέσκα, Λέω για άλλε χώρε. Άλλες. Και σε κάποιε άλλε χώρε, αντιθέτω, θα πρέπει κανείς να τα λέει με έναν τρόπο συμπαθητικό, προσεκτικό, έτσι, όπως κάνουν οι Κινέζοι και οι Ιαπωνέζοι. Ε, Επομένω, εμεί τριζόμαστε πάνω σα, τόσο ώστε να μπορέσετε να βρείτε την κατάλληλη διατύπωση. James Ellis. Euh, δεν ξέρω, δεν ξέρω, Πρόεδρε, λέει ο κύριο Έλλη. Σήμερα το πρωί διαπίστωσα ότι εδώ οι φίλοι Γεωργίου Τραπέζη, ο Φερνάντε μίλησε στα αγγλικά, ένα και εγώ Άγγλο μου μιλήσω στα γαλλικά, όμως έτσι θα μπερδέψω του. Τέλος πάντων. Εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής. Όχι, δεν είναι δυνατόν να παραβλέπουμε ότι το κλίμα είναι κλίμα λιτότητας στις χώρες μας. Οπότε, όσον αφορά τώρα τον προϋπολογισμό, θα πρέπει να προσέξουμε μην στείλουμε το λάθος μήνυμα. Γιατί πέφτουν φόροι παντού στη χώρα μας. Και να πούμε εμείς ότι δεν θα κάνουν προβλησμό λιτότητας, ίσως δεν είναι και το πιο καλό. Άρα, να πιάσουν τόπο τα, τα λεφτά και υπόριο. Βάλει φορμάνι. Και βλέπω εδώ πέρα το σχετικό κομμάτι στο κείμενο και, και ακριβώ όπω ελέγχθη, θα πρέπει να κάτσουμε και να μελετήσουμε όλες τις δραστηριότητε και, και να δούμε αν πραγματικά χρειάζεται να τηρήσουμε όλες τις υποχρεώσεις που έχουμε δεσμευτεί να τηρήσουμε. Για να σας τα πω στα αγγλικά τώρα. Να συρρυκνώσουμε τις δεσμεύσεις, οι υποχρεώσεις, ώστε να συρρυκνωθούν και τα ράλα, αντίθετα τα υπόλοιπα προς εκαθάριση και έτσι να κάτσουμε στα γαλλικά τώρα να δούμε θα γίνει με όλα αυτά τα κονδύλια που χρειαζόμαστε και να, να, να, να δούμε πώς η η κακή εκτέλεση φετινή να μην παντού το 2012. Γιατί θα πρέπει πραγματικά να αξιοποιήσουμε το, το, το, κάθε δεκάρο, το κάθε ευρώ που έχουμε στη μα. Επίση, ε, όσον αφορά τη στρατηγική το 2020, θα πρέπει επίση να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε. Και από την άλλη μεριά, δεν χρειάζεται για όλε τι δραστηριότητε του 2020 ε, χρήμα. Όμως θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αυτή η απορρίθμιση. Χρειάζεται ανάληψη δράση στα κρατημέλη και όχι αναγκαστικά περισσότερα χρήματα. Τώρα όσον αφορά την ε, διατύπωση συμφωνώ με τον κύριο Ραγκλίνο ότι είναι κάπως έντονη η διατύπωση. Λέει ότι δεν οποιαδήποτε προσπάθεια να συρρυκνώσει τον προπολογισμό θα είναι πάρα πολύ καταστροφικό για την Ευρωπαϊκή Ελληνική. Αυτό είναι πάρα πολύ έντονο, ακραίο. Ναι, παντού έχουν παγώσει οι προπολογισμοί. Αλλού έχουμε περικοπές στον προπολογισμό. Προσοχή γιατί έχουμε και το, την προπονή του 2012 που θα, πρέπει να αναδείξει, να τονίσει αυτό το οποίο κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάμε μπροστά. Αλλά επίση θα πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι και εμεί δεν είμαστε αυτοί που θέλουν να ξοδέψουν περισσότερα. Αυτό δεν μπορεί να περάσει στην Αγγλία με τίποτα. Bien, merci James. Monsieur Portage. Ευχαριστούμε ο κύριος Πόρτας. Il s'est couvert de gloire dans Commission Chour, euh, dans son débat avec... Εδώ είναι πολύ ένδοξη ημέρα γιατί σα θυμίζω και τη συζήτηση με τον κύριο Λεβαντόσκη. Δεν ξέρω αν ε, είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλοι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ότι εδώ αν το μόνο πρόβλημα του εγγράφου ήταν γλαισίκο, όλα θα είχαν λυθεί. Νομίζω ότι το πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας και το λέω ειδικό στην ε, κυρία Μπαλτζάνη, είναι το πρόβλημα μιας ε, αντίφασης ασυμβίβαστης. Διότι εδώ νομίζω η συγγήτρια είναι πεπισμένη ότι ο ευρωπαϊκός προπολογισμός πρέπει να ε, χρησιμοποιείται, να χρησιμεύει για τη δημιουργία απασχόλησης, για να στηρίζει μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης. Και Βεβαίω πρέπει ο ευρωπαϊκό προπολογισμό να υπάρχει μαζί με του εθνικού προπολογισμού. Όμω το σημερινό τοπίο αυτό που συμβαίνει είναι ότι θα έχουμε ένα προπολογισμό με μηδενική αύξηση. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα, θα είχαμε πραγματικά ανάπτυξη αν μπορούσαμε να αφαιρέσουμε την, τον πληθωρισμό. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα τώρα. Μπορούμε να αρχίσουμε να συζητούμε αν η στατιακή 2020 είναι χρήσιμη για κάτι ή για τίποτε. Όμω, κατά τη δική μου άποψη, για πολύ λίγα θα χρησιμεύσει. Διότι είναι πάρα πολύ ωραίε και ευχάριστε ε, δηλώσει αυτή στατικική. Εδώ λοιπόν έχουμε μια άποψη κάπως διαφορετική από τη συναδέλφου Βαλτζάνη. Ίσως θα μπορούσε το θέμα να επιληθεί εάν διερευνούσαμε όλες τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού και Εθνικών προπολογισμών. Η μόνη όμω σχέση συνεργασία που μπορώ εγώ να διαδώ ε, μεταξύ ευρωπαϊκού προπολογισμού για το 2012 και των μελλοντικών προπολογισμών ε, για το 2012 της κάθε χώρας, η μόνη δυνατότητα συνεργασίας που βλέπω εγώ είναι η μείωση των δαπανών. Δεν βλέπω καμία δυνατότητα πρακτικότερης συνεργασίας. Πρέπει να μειώσουμε, να μειώσουμε και να ξαναμειώσουμε τις δημόσιες δαπάνες. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι το τοπίο στο οποίο βρισκόμαστε. Δεν βλέπω άλλες δυνατότητες συνεργασίας. Άρα, προφανώς είμαι υπέρ του σωστού εντοπισμού των αρνητικών προτεραιοτήτων ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Και χρειάζεται μια πολύ καλή μελέτη των δυνατοτήτων ε, ευελιξίας. Εδώ συμφωνώ απολύτω. Δεν έχω όμω αυταπάτε δεν έχω μεγάλες αυταπάτες γενικότερα πλέον για το ευρωπαϊκό εξάμεινο, όπως ε, έχει περιγραφεί. Εγώ δεν έχω καμία τέτοια ψευδέστηση ότι θα μας επιτρέψει καλύτερο, καλύτερο συντονισμό των πολιτικών ε, αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Όπως έχει ε, ξεκινήσει αυτή τη χρονιά, όπως έχει περιγραφεί, έχει έναν και μοναδικό στόχο. Λιτότητα, λιτότητα και ξανά λιτότητα. Ε, αυτό το λέω προ του αγαπητού σα συναδέλφου. Είτε αυτή την γνωμοδότηση είτε με όλου. Άλλη λιτότητα παραπάνω δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Certes. Αν κανεί δεν έχει νερό, πώ να ποτίσει όμω. Αυτό είναι το πρόβλημα φέτο. Ιζαμπέλ Τυρό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστούμε την ε, εισηγήτρια με την οποία συμφωνούμε. Προσυπογράφουμε την γραμμή πλεύσης που εχάραξε και για σταδιακή 2020 και για το ότι χρειάζεται να δημιουργηθούν θέσει εργασία. Συμφωνούμε σε όλα αυτά που είπε. Ακριβώ πρόκειται για μια λιτότητα που έχει επιβληθεί σε όλου. Όμω αυτό δεν αποτελεί όραμα, σχέδιο πολιτικό. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να δημιουργήσει κανεί απασχόληση και επομένω η λιτότητα πάλι είναι ένα κομμάτι της διαδρομής. Δεν μπορεί αυτό να είναι το πνεύμα που διαπνέει τον προϋπολογισμό. Οπότε, ε, έτσι όπως ακριβώς είναι η κατάσταση, δεν νομίζω θα πρέπει σε αυτό το προϋπολογισμό να έχουμε ε, κάποιες σκέψεις για το τι γίνεται σήμερα. Στο κείμενό σας μάλλον έχουμε ε, κάτι, κάποιο σχόλιο για, το αυτό, που γίνεται στον αραβικό κόσμο, χωρίς να καθόμαστε να βλέπουμε σημείο προς σημείο, να, να, να διαπιστωθεί ότι είναι πάρα πολύ αποφασιστικό, κρίσιμο, καθοριστικό αυτό που γίνεται σήμερα. Οπότε κάτι πείτε στο ψήφισμά σας. Ο Πρόεδρος, Ιζαμπέλ, σε ευχαριστούμε. Ναι, ναι, νομίζω ότι εγγράφω σε αυτό να τα πούμε, να τα πεις τέλος πάντων στην συγκήτρια, θα την ενδιαφέρει με Γκόραν Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και εγώ από τον Βορρά θα πάει, ήθελα να πω ότι στην Φιλανδία υπάρχει ανοιχτό όμως τόνο στην πολιτική συζήτηση σίγουρα. Ίσως όμω ε, η διαφοροποίηση είναι σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία μια και το αντευρωπαϊκό κόμμα είναι το πιο γοργά αναπτυσσόμενο στη Φιλανδία τώρα. Δεν αντέδρασα ουσιαστικά όπως ε, ο συνάδελφος διότι ήταν διπλωματική πίστευα η Φραντσέσκα στο εγγραφό της ε, στις διατυπώσεις της παρόλα αυτά συμφωνώ με τον Χάρλ δεν υπάρχει λόγος να έχουμε μεγάλες αντιπαραθέσεις για τις διατυπώσεις ή να είμαστε προκλητικοί σε σχέση με αυτές τις διατυπώσεις πρέπει να επικεντρωνόμαστε στην ουσία και όχι με κάποιες άλλες ε, υπερβολές και για τη διατύπωση αυτό εντάξει τώρα για την ουσία νομίζω είναι τεράστια σημασία να πούμε όπως είπε η κυρία Ντουιρόν, ότι πρέπει κάτι να κάνουμε επιτέλους για αυτά τα οποία θεωρούμε ότι είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό πάνω από την επικέντρωση που επέλεξε η Φραντσέσκα για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τις επενδύσεις, δεν θα ήθελα να καταθέσω τροπολογίες στις διάφορες κατηγορίες ή στα διάφορα κονδύλια θα ήθελα να πόσχω από αυτό. Είναι πολύ καλό ότι ήταν σύντομη η Φραντσέσκα και στοχοθετημένη. Να μην περάσουμε στι επιμέρου κατηγορίε και κονδύλια. Απευθύνω έκκληση στι άλλε κοινοβουλευτικέ ομάδε και κοινοβουλευτικέ επιτροπέ να μην καταθέσουν τροπολογίε, ώστε να, είναι, να μην έχουμε ένα μεγάλο εύρο ε, για τι διάφορε κατηγορίε και κονδύλια. Πρέπει νομίζω όμως να κρατήσουμε τις αρχές για τις οποίες δώσαμε αγώνα πέρυσι και να τις διατηρήσουμε. Η ομάδα μου κάποιες τροπολογίες θα καταθέσει, μία ή δύο δεν ε, το έχω υπόψη ακριβώς. Αλλά σε σχέση με τη σπουδαιότητα, τη σημασία που θα μπορέσει να δοθεί στην, στον προπολογισμό για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσει που έκανε λόγο η Φραντσέσκα για τι θέσει απασχόληση, τι αντιμετωπίσει των προκλήσεων κτλ. Κάποιες τροπολογίες λοιπόν όπως είπα θα καταθέσουμε, αλλά γενικότερα για την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις και όχι στι επιμέρους κατηγορίες ή κονδύλια. Αυτό είναι σημαντικό. Ευχαριστώ. Merci, Göran. Ε, Ευχαριστούμε, Γκέραν. Απλώς και εγώ θα στηρίξω αυτήν την ε, φιλοσοφία της όλης αυτής διαδικασίας των κατευθυντηρίων γραμμών. Σωστά την ακολουθεί η κονδυλια αυτο ειναι σημαντικο ευχαριστω merci ευχαριστουμε γκεραν απλως και εγω θα στηριξω αυτην την φιλοσοφια της ολης αυτης διαδικασιας των κατευθυντηριων γραμμων σωστα την ακολούθη η συγκεντριά μας. Και σωστά το υπογραμμίζετε κι εσείς. Εδώ επίσης να υποσημειώσω ότι υπάρχει εδώ μια σημαντική ενοιολογική απόχρωση. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ Σουηδικών των Σουηδών και Σουηδικών των Σουηδόφωνων Φιλανδών, στον τρόπο που εκφράζονται. Προφανώς ε, οι γλωσσικές αυτές αποχρώσεις θα είναι ακόμη πιο εύγλωτες μετά από τις όλες ε, συζητήσεις μας σήμερα. Κυρία Αντρέασεν, τελευταίο ομιλητρία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να επαναλάβω τα επιχειρήματα τα οποία είχα παρουσιάσει όταν βρισκόμαστε στην ίδια φάση των διαπραγματεύσεων σε σχέση με τον περιβολισμό του 2011 θα έλεγα ότι αυτό εδώ το Ευρωκοινοβούλιο και σε γενικότερους όρους η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχής στις ε, δημοσιονομικές αυτές, ε, στα δημοσιονομικά εγχειρήματα ή τον προπολογισμό και αυτό είναι εξόφθαλμο με τις μεταφορές που ζητείτε να εγκριθούν κάθε χρόνο και με τα μη, ε, εξοφλη, μη τα πανηθέντα κατά τα τέλη ενός έτους από πλευράς κονδυλίων. Πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια λοιπόν να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην χρήση των κονδυλίων σε σχέση με τον προϋπολογισμό και δεν προβλέπω σε αυτό το εγχείρημα ότι θα υπάρξει κάποιο περιθώριο για αυξήσει. Και επιπλέον κιόλα υπάρχει περιθώριο μειώσεων στον προπολογισμό υπό πραγματικού όρου. Το άλλο θέμα που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι η στρατηγική για να διεξέλθουμε από την κρίση δεν είναι η στρατηγική της Ευρώπης του 2020. Η στρατηγική για την έξοδο αυτή Ίσως θα έπρεπε να είχε ήδη δομολογηθεί και θα έπρεπε ίσως να ήταν η στρατηγική για τη Λισαβόνα. Σε σχέση με αυτό το έγγραφο λοιπόν από πλευρά Φραντσέσκα για την αναφορά για την Λισαβόνα και την στρατηγική του 2020, δεν είναι ακριβώς το θέμα της ζήτηση ε, νέων κονδυλίων. Αυτό δεν μας καθιστά ιδιαίτερα αξιόπιστος. Θα πρέπει να μας προβληματίσει αυτό λίγο παραπάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, Φραντσέσκα, Θέλετε να κάνετε κάποια καταληκτικά σχόλια για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ. <clears throat> Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους. Νομίζω ότι συμφωνούμε ως προς την ιδέα να επικεντρωθούμε σε σημαντικά θέματα. Κυρίως να δώσουμε μεγάλη έμφαση στη στρατηγική του 2020. Θυμίζω ότι ο ορισμός των τομεακών προτεραιοτήτων θα πρέπει να γίνει με την συμμετοχή των ειδικευμένων αρμόδιων επιτροπών. Θυμίζω ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή τη διαδικασία του προπολογισμού, τη στιγμή που ορίζουμε τι κατευθυντηρίε γραμμέ. Έπειτα θα πρέπει να περάσουμε και σε ένα ακόμη πιο ευαίσθητο θέμα. Δηλαδή να δούμε του αριθμού, τα αριθμητικά στοιχεία. Εκεί θα μπορέσουμε πιο συγκεκριμένα, πιο πρακτικά να εντοπίσουμε πολιτικέ προτεραιότητε. Ε, ως προς αυτό, επειδή βλέπω ότι επέστρεψε σήμερα το ζήτημα επιτάπητος, είναι το τι θα κάνουμε ακριβώς με τις αρνητικές προτεραιότητες. Θυμίζω εδώ το εξή. Μπορεί τελικά να καταλήξουμε ότι δεν έχουμε και αρνητικέ προτεραιότητε, διότι είναι ιδιαίτερα περιορισμένος ο μας μα. Ε, εδώ σίγουρα θα φροντίσουμε να έχουμε μια πολύ, μια πολύ καθορισμένη, αυστηρά καθορισμένη μέθοδο, αλλά ελπίζω όλοι να κάνετε και πολύ συγκεκριμένε πρακτικέ προτάσει ώστε να μπορέσουμε να δούμε ποιε είναι οι αρνητικέ προτεραιότητε. Ε, έπειτα, ε, σα εγγυώμαι ότι θα συζητήσω με τι ε, ειδικέ επιτροπέ, ώστε να έχουμε και μια πιο επίσημη, πιο έγκυρη πολιτική συζήτηση και να καταλήξουμε και για το σχέδιο προπολογισμού που θα μα φτάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη Απριλίου. Και έπειτα θα έχουμε να λάβουμε και μια απόφαση για το σχέδιο αυτό προπολογισμού στι αρχέ Μαΐου τότε θα μπορούμε ακριβώς να καθορίσουμε και κάποιες γραμμές συγκεκριμένε, κάποια όρια για τις τομεακές πολιτικές σε συνεργασία με αυτές τις ειδικέ επιτροπές και να παραμείνουμε, να μείνουμε μάλλον και πιο, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι στα αριθμητικά στοιχεία. Φέτος, όπως έχω πει, θα πρέπει να δούμε μια πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάπως διαφορετική από ό,τι φανταζόμαστε συνήθω και σε σχέση με τον δημοσιονομικό ε, προγραμματισμό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Φραντζέσκα, ευχαριστούμε όσους έλαβαν το λόγο. Να θυμίσω ότι για το σημείο αυτό, για την έκθεση αυτή, διαπιστώσαμε και αποφασίσαμε στη συνεδρίασή μας στις 7 Φεβρουαρίου, λόγω των προθεσμιών, να μην σεβαστούμε δυστυχώς τις κλασικές προθεσμίες για μετάφραση. Οι τροπολογίες λοιπόν πρέπει να υποβληθούν πριν τις 8 Μαρτίου το μεσημέρι στα αγγλικά. Αυτό ούτως ή άλλως θα διευθετήσει και το πρόβλημα των συνδικών. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Δεν θα δούμε αυτή τη στιγμή το σημείο 5 που αφορά ειδικά τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου ακριβώς λόγω των όσων υπόθηκαν προηγουμένω από τον κύριο Φερνάντε, Θα επανέλθουμε αργότερα. Σας προτείνω να περάσουμε τώρα στο σημείο 20 με εισηγήτρια την κυρία Τρίπελ. Θα μας παρουσιάσει αρκετές τροπολογίες σήμερα αλλά θα ήθελα να δούμε τώρα συγκεκριμένα τη χρηματοδότηση τη υπηρεσία εξωτερικής δράση με την κυρία Τρούπελ, όπου ο ε, οικονομικός διευθυντής της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης βρίσκεται μαζί μα. Επειδή ο κύριος Άκμοντ επίσης θέλει να συζητήσουμε το δικό του σημείο ακριβώ μετά, θα ήθελα αυτή τη στιγμή να δούμε συγκεκριμένα τη χρηματοδότηση της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, να ψηφίσουμε και μετά βλέπουμε το σημείο κ. και να μπορέσουν όλοι οι συνάδελφοι να ακολουθήσουν το πρόγραμμα που θέλουν. Κυρία Τρίπελ, θα μας παρουσιάσετε το θέμα αυτό. Okay, thanks, um, Allah. Ευχαριστώ, αλλά το EAS έχει υποβάλει αίτηση μεταφοράς για τα κεφάλαια μεταξύ των γραμμών για την ασφάλεια και την εποπτεία και τις άλλες ε, λειτουργικές δαπάνες. Δαπάνες σε σχέση με τη διοργανική συνεργασία για 1,6 συνολικά άθροισμα εκατομμύριων ευρώ. Λέγεται ότι χρειάζονται αυτά τα κονδύλια ως επιχείρημα για να μπορούν να προσλάβουν εξωτερικούς υπαλλήλους ώστε να προπαρασκευαστεί η διαχείριση ενός ε, νέου, σε σχέση με ένα νέο κτίριο του EASS. Και έτσι λέγεται ότι θα υπάρξει το Service Level Arrangement μεταξύ του EAS και των ανθρώπινων πόρων, ανθρώπινων δυναμικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση επίσης και για τις υποδομές και τα κτίρια. Για να σας δώσω μια πρώτη, ας το πω έτσι, γεύση της θέσης μου σε σχέση με τα σχόλια σχετικά, εγώ εκφράζω κάποιες αμφιβολίες για το γεγονός ότι οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τον προϋπολογισμό του EAAS και θα ήθελα επεξηγήσεις από το EAAS. Δεν θα ήταν πιο σωστό αυτοί να πληρώνονται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νομίζω ότι θα ήθελα να έχω περισσότερες πληροφορίες όπως και άλλοι ευρωβουλευτές για το service level arrangements, τις ε, συμβατικές υποχρεώσεις για τέτοιου είδους υπηρεσίες. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων ευρωβουλευτών και θα επανέλθω με τη σύστασή μου. Ευχαριστώ. Je Σας ευχαριστούμε. Δεν ζητεί κανένα συνάδελφο το λόγο. Ίσως λοιπόν ο κ. Τσάιλ δεν θέλει να απαντήσει απευθείας στην ερώτηση της εισηγήτριας. Διευθυντά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι είμαστε σχετικά νέοι σε σχέση με αυτή τη διαδικασία διαχείρισης των κονδυλίων του προπερισμού μας και είναι μια καλή ευκαιρία για μας έτσι να μπορέσουμε να συμμεριστούμε τον προβληματισμό μας με την δική σας κοινοβουλευτική επιτροπή. Αυτή η συγκεκριμένη μεταφορά, όπως είπε η συγκήτρια, στοχεύει στο να μπορέσουμε εμείς στο τέλος να καταφέρουμε να πληρώσουμε για κάποιες υπηρεσίες που μας παρέχονται από διαφορετικά τμήματα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να βοηθηθεί η υποστήριξη, η συνδρομή, η διοικητική για τους υπαλλήλους μας από πλευράς υπαλλήλων, ιδιαίτερα σε σχέση με εκείνους που έχουν προσθεθεί στην εξωτερική υπηρεσία από την Γραμματεία του Συμβουλίου και που προηγούμενα ήταν υποδιαχείριση για την πληρωμή των μισθών τους και άλλων παροχών που τους δίνονται μέσω των άμεσων υπηρεσιών του Συμβουλίου διοικητικά. Και τώρα που ζητήθηκε η, η Ευρωπαϊκή υπηρεσία, η Επιτροπή με τι υπηρεσίε τη να καλύπτει αυτέ τι δαπάνε, πρέπει να εξοφληθούν αυτέ στην Επιτροπή. Είναι τεράστια, α το πω έτσι, η εμβέλεια αυτή ε, του οργανικού συσχετισμού σε σχέση με το e για να μπορέσει να δημιουργηθεί η δυνατότητα πρόσθετων υπηρεσιών όταν αυτό μπορεί να παρέχεται από τα όργανα, τα θεσμικά όργανα και έτσι να υποφεληθούμε από τις οικονομίες κλίμακος. Ο στόχος τώρα είναι να διασφαλίσουμε ότι στα αντίστοιχα κονδύλια για τη διοργανική συνεργασία θα έχουμε επαρκή κονδύλια, επαρκή ποσά για να καλύπτονται οι αναμενόμενες δαπάνες <clears throat> για την πλήρη στελέχωση από πλευρά υπαλλήλων για την υπηρεσία εξωτερικών ε, δράσεων προτείνουμε να πάρουμε χρήματα από ένα κονδύλιο ε, μεταφοράς όσον αφορά την ασφάλεια για, την, για τα κτίρια και την εποπτεία. Δεν αναμένεται ότι θα χρειαστεί το πλήρε ποσό για το νέο κτίριο, γιατί κατά το τέλειο του θα μετακινηθούμε. Αλλά ε, όπω φαίνονται τα πράγματα σήμερα, μπορούμε ήδη να πούμε ότι υπάρχει ήδη κάποιο ε, πλεόνασμα. Ο στόχο, όπω είπα, το νόημα του εγχειρήματο είναι να διασφαλίσουμε ότι θα είμαστε σε θέση να, ανταποκριθούμε στι υποχρεώσει που έχουμε συμβατικά να λάβει με τα άλλα θεσμικά όργανα, ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνδρομή αυτή. Δεν θα ήταν αποτελεσματικό σε σχέση με την υπηρεσία αυτή να δημιουργηθούν προβλήματα, αλλά σε σχέση με τι πρόσθετε δαπάνε που συμφώνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλύπτει σε σχέση με εμά και με τα νέα στελέχη που θα προσέρχονται στο EAAS από τη Γραμματεία του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Merci. Ε, σας ευχαριστώ. Για να είμαι βέβαιος ότι κατάλαβα σωστά, αυτού του είδους η χρηματοδότηση, η πληρωμή, είναι κάτι που το χρειάζεστε τώρα. Διότι είναι η πρώτη χρονιά κατά την οποία λειτουργεί η υπηρεσία σας. Πρέπει να μεταφορθεί λοιπόν αυτή η πληρωμή προς την υπηρεσία εξωτερικής δράσης από από τι βασικές υπηρεσίες προσωπικού, ιδίω τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φαντάζομαι από του χρόνου δεν θα έχετε ανάγκη τέτοιου είδους ε, συσχετισμό λογιστικό μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή δράση και φαντάζομαι Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σωστά είναι μια και έξω, αν μπορώ να το πω έτσι. Συμφωνώ μαζί σα Πρόεδρε, ότι κατά τη διάρκεια αυτή τη ας το πω έτσι, πρώτης πρώτη ε, φάσης στα σπάργανα ακόμα, ε, αυτό θα είναι πιο αναγκαίο ε, περισσότερο, μια και οι συμφωνίε συμβατικά που έχουμε συνάψει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Γραμματεία του Συμβουλίου ολοκληρώθηκαν μόνο κατά το ύστερο τμήμα τη περσινής χρονιά και μετά από την την, τον καθορισμό τη δομή του προπολογισμού προηγούμενα και στου επόμενου προπολογισμού θα προσπαθήσουμε να είμαστε πιο επακριβείς προβλέποντας τι πραγματικέ δαπάνε στα διαφορετικά κεφάλαια και θα χρειάζονται λιγότερο τέτοιου είδου προσαρμογέ μεταξύ των διαφορετικών κεφαλαίων στο μέλλον, στον προπολογισμό. Ευχαριστώ. Ο κύριο Πόρτα, παρακαλώ, ζήτησε τον λόγο. Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Αν το σύνολο αυτών των έξι μεταφορών εδώ, αν αντανακλάται σε αυτό το σημείο και βρίσκεται αυτό συνολικά συζήτηση κυρίως επειδή υπάρχει μία μεταφορά για την οποία θα ήθελα να παρέμβω εγώ σχετικά και είναι η μεταφορά 1.500 ευρώ μηνιαία για την, ε, τα θέματα των ε, βουλευτών και των ε, βοηθών τους. Αυτά δεν βρίσκονται υπό έτσι και δεν θα ψηφιστούν σήμερα. Έτσι θα ακολουθήσει αυτό. Λοιπόν, για το σημείο 20. Το ρωτάω αυτό. Πότε θα συζητηθεί και πότε θα αποφασιστεί αυτό. Ευχαριστώ. Αργότερα. Εντάξει, πλούτα. Δεν ζητεί άλλο το λόγο. Εισηγήτρια, η δική σας άποψη. Um, η κυρία Τρίπερ. Λοιπόν, δεδομένου του γενικότερου συμφέροντο και ενδιαφέροντο να δημιουργηθεί αυτό το νέο EAAS, θα ήμουν υπέρ αυτή τη μεταφορά, λοιπόν τελικά. Ευχαριστώ. Υπέρ. Σα ευχαριστούμε. Ψηφίζουμε λοιπόν για αυτήν την μεταφορά, μόνον αυτή τη μεταφορά. Αργότερα θα δούμε άλλε τη συζητητριά μα. Ποιο είναι υπέρ τη μεταφορά αυτή. Ευχαριστώ. Κατά. Μία ψήφο κατά. Αποχές. Δεν υπάρχουν αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν με ευρία πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε πλέον να περάσουμε. Θα επανέλθουμε, θα επανέλθουμε στις υπόλοιπες ε, Μεταφορέ τη κυρία Τρούπελ αργότερα. Όμω τώρα θα έλεγα να περάσουμε στι δύο εκθέσει που θα μα παρουσιάσει εντάχει ο συνάδελφο Άγμον. Πρώτα απ' όλα, αντικαθιστώντα την κυρία Γένσεν, που δυστυχώ δεν θα έχουμε τη χαρά να ε, βλέπουμε μαζί μα σήμερα και έπειτα τη δική του. Πρώτα λοιπόν για το μέλλον της δημοσιονομικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σημείο 11. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για αυτή την ευελιξία σε σχέση με το πρόγραμμα. Είναι μια γνωμοδότηση της κυρίας Γένσεν που δυστυχώς δεν μπορεί να παραστεί σήμερα. Συνέταξε μια ενδιαφέρουσα γνωμοδότηση που απλά και μόνο αναφέρεται στις επικρίσεις που είχαν ασκηθεί σε σχέση με αυτόν τον σχετικά νέο τρόπο να εργαζόμαστε για την πολιτική για την ανάπτυξη όπου κυρίως εξετάζονται από πλευρά τη τα σημεία εκείνα τα οποία είχε θίξει το ελεγκτικό συνέδριο που είχε συντάξει μια πολύ επικριτική έκθεση και αναφέρεται σε κάποια θέματα που θα ήταν χρήσιμο να τύχουν συνέχεια και να σχολιαστούν. Υπογραμμίζει επίση το γεγονό ότι δεν μπορούμε ισοπεδωτικά με μια προσέγγιση να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα όπω ε, συμβαίνει και με την Επιτροπή και επιθυμεί να τα υπογραμμίσει αυτά τα θέματα. Χρειάζεται επίση ένα υγιέ πλαίσιο διαχείριση αυτό πρέπει ακόμα να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί στη συνέχεια μετά. Επίσης υπογραμμίζει το γεγονός ότι θα έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερη συνειδητοποίηση σε σχέση με τι χώρε μα μας και με τους χορηγούς αλλά και με τις ε, χώρες αποδέκτες για να δούμε τι γίνεται σε σχέση με αυτό το μέσο και ποια είναι τα αποτελέσματα τελικά ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία σε σχέση με τους πολίτες ε, για τις προσπάθειες να επωφεληθούν αυτές οι χώρες από αυτές τις δράσεις. Μετά υπάρχει η εκτενέστερη ευρύτερη συζήτηση σε σχέση με την ε, αντανάκλαση στον προϋπολογισμό από τις νέες, ε, για τις νέες αυτές τα, ανάγκες με ένα πολύ ισορροπημένο τρόπο γίνεται αυτό λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό και θεσμικό σκηνικό και τα προηγούμενα ιστορικά τα οποία μας οδήγησαν στην κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα και εν κατακλείδη τέλος υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος συντονισμός ε, σε σχέση με το σεβασμό των υποχρεώσεων από πλευρά ε, προπολογισμού εναντί τρίτων χωρών. Να αποφύγουμε επικάλυψη πολιτικών όπως συμβαίνει πολλές φορές σήμερα. Και ταυτόχρονα τονίζει το γεγονός ότι επίσης θα έπρεπε να υπάρξει προβληματισμός που μπορούμε να υπο, ε, ευθυγραμμίσουμε τις ανάγκες μας ε, και τις υποχρεώσεις μας σε σχέση με τις ανάγκες αυτών των χωρών. Υπάρχουν διαφορετικές ε, αιτήσει και ανάγκες σε σχέση και με τα διάφορα κράτη. Αυτά όλα αντανακλώνται στην γνωμοδότηση της κυρίας Γένσεν συνολικά. Θα, όπως αναφέραμε δεν μπορεί να παραστεί και αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Nous préparons une réponse du Parlement Πρόκειται για μια απάντηση λοιπόν της Ευρωπαϊκής ε, σε μια πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απάντηση του Κοινοβουλίου σε αυτά. Εξ ονόματός μου θα ήθελα να πω ότι βλέποντας ε, τις σημαντικές αλλαγές και μεταβολές και όλα όσα έχουν συμβεί στη νότια όχθη της Μεσογείου θα πρέπει να οδηγηθούμε στο να ξαναπροβληματιστούμε τους όρους ε, τους οποίους παρέχουμε αυτή τη βοήθεια ο επόμενο αγορητής. Έχω κάποια σχόλια για αυτά τα θέματα. Ουσιαστικά συμφωνούμε με την κυρία Γένσεν σε αυτά που λέει. Δηλαδή με άλλα λόγια για την βασι... τον βασικό προσανατολισμό της γνωμοδότησής της που είναι καλός. Κάποια πράγματα θέλουμε να δούμε και να θα καταθέσουμε ίσως και κάποιες τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να τονίσουμε κάπως περισσότερο ότι η συνδρομή από πλευράς προϋπολογισμού με κονδύλια είναι ένα σημαντικό και καλό μέσο που θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερο ρόλο να διαδραματίσει στην πολιτική για την ανάπτυξη από ό,τι έχει μέχρι σήμερα. Και αυτό για πολλούς και καλούς λόγους. Είναι ένα μη γραφειοκρατικό μέσο. Αν μπορούμε να έχουμε το, τα σωστά μέσα και εργαλεία για την στάθμιση και αξιολόγηση των αναγκών και όταν θέλουμε να βελτιωθεί ε, το δυναμικό και η ικανότητα για εκδημοκρατισμό πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πιο επακριβείς όταν έρχεται η ώρα για σαφείς συντελεστές για να έχουμε μια καλή αξιολόγηση τέτοιου είδους συνδρομής με κονδύλια με σαφείς προσδιορισμούς και μια ε, εκτενή ε, εποπτεία, σαφή εποπτεία, ώστε να αποφύγουμε προβλήματα. Τρίτον, η κυρία Γένσεν αναφέρει την ανάγκη να εμπλακεί η κοινωνία των πολιτών, η δημοκρατική κοινωνία εδώ. Και εδώ πρέπει να είμαστε πιο σαφείς και ε, ξεκάθαροι για να είναι διαφανής αυτή η διαδικασία και να μην είναι στα χέρια της διακυβερνητικής διαδικασίας συστηματική εμπλοκή των κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών στο διάλογο για τα θέματα της ανάπτυξης και μέσω αυτών των μέσων και εργαλείων. Και τέλος, είναι σημαντικό να, αυξήσει, αυξηθεί ο συντονισμός μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πραγματική δύναμη στην Ευρωπαϊκή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγαλύτερο βάρος συνολικά από ότι τα επιμέρους κράτη-μέλη. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειωθεί το γραφειοκρατικό βάρος, όχι μόνο στις χώρες μας, αλλά και στις χώρες αποδέκτες θα έπρεπε να θέσουμε μεγαλύτερο βάρος στο συντονισμό και σε σχέση και με αυτό το μέσο μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταφέρουμε τέλος να έχουμε περισσότερα αποτελέσματα, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί με τη σύνδρομη αυτή, με τα κονδύλια που διαθέτουμε. Θα καταθέσουμε κάποιε τροπολογίε για αυτά τα θέματα, αλλά ουσιαστικά συμφωνούμε για την κατεύθυνση αυτή τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Merci, ε, Ευχαριστούμε, Γκέραν. Η συντονία η οποία θα μιλήσει εξ ονόματο ε, του ε, συναδέλφου του ΕΛΚ για το θέμα αυτό. σε ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω μια επιστολή μπροστά μου από τον συνάδελφο Κοσλόφσκι που θα σας διαβάσω και για την ε, ευθύνη για αυτή τη νομοδότηση. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λυπούμε πολύ λόγω του γεγονότος ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Ζάγκρεπ και συμμετέχω σε μια συνεδρίαση του Προεδρείου του ΕΛΚ, δεν είμαι και δεν θα είμαι σε θέση να παραστώ ανάμεσά σας να συζητήσω τη συνδρομή στο μέλλον για τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, εγώ ίδιος. Στην αρχή αυτής της επιστολής θα ήθελα να διασφαλίσω να σας ε, εγγυηθώ για το σεβασμό μου και να συγχαρώ την εισηγήτρια για τη γνωμοδότηση, τη συντάκτρια γνωμοδότηση. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η γνωμοδότηση και είναι πολύ καλά στοχοθετημένη και έχει ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με την Επιτροπή Προπολογισμών. Θα έλεγα ότι το θέμα τη εγγραφή στο προπολογισμό των μέσων για την ανάπτυξη είναι πολύ μεγάλη σημασία ε, όταν βρίσκεται εκτός ε, ελέγχου και καθορισμού του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου είναι ε, επιζήμιο και για την πολιτική για την ανάπτυξη αλλά και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιζήμιο. Θα πρέπει λοιπόν να εντάσσεται στον προπολογισμό. Όσον αφορά τι τροπολογίε, θα ήθελα να αναφέρω ότι θα είναι συμπληρωματικέ αυτέ οι τροπολογίε και δεν θα έχουν μείζωνα επίπτωση όσον αφορά τις προτάσεις που υποβάλλει η συντάκτρια της Η παραγωγικότητα θα έλεγα της ε, πολιτικής για την ανάπτυξη έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό, διότι ιδιαίτερα συχνά η συνδρομή από πλευράς προϋπολογισμού με τα κονδύλια αυτά διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο και για τους εθνικούς προϋπολογισμούς των αναπτυσσόμενων χωρών. Γι' αυτό θα, θέλα θα έπρεπε οι αναπτυσσόμενες χώρες να συντάσσουν ε, τα δικά τους, να καταρτίζουν τα δικά τους σχέδια με δικές τους προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα μέσα και τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η συνδρομή που τους δίνουμε από πλευράς κονδυλίων θα έπρεπε να έχει μια φύση πολιετούς χαρακτήρα, ε, να γίνεται ε, σε ένα πολιτές πλαίσιο. Και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καλύτερο συντονισμό σε σχέση με αυτό το έργο και θα πρέπει να επιμερίζουν το έργο και τις αρμοδιότητες. Αυτό είναι το ε, νόημα και της Task Force για την αποτελεσματικότητα, διότι όταν υπάρχουν επικαλύψεις ή όταν υπάρχει για παράδειγμα έλλειψη, απουσία συνεκτικότητας και συνοχής σε αυτές τις δράσεις, υπάρχουν προβλήματα προβλήματα τα οποία ε, ανακύπτουν και τα οποία αναφέρει και η συντάκτρια νομοδότηση στην έκθεσή τη. Η συνδρομή μα από πλευρά κονδυλίων, από πλευρά προπολογισμού είναι τόσο σημαντική που γι' αυτό είναι σημαντικό να υπογραμμιστούν εδώ τα θέματα τα οποία αναφέρω στην επιστολή μου. Ευχαριστώ. Σα um, Σας ευχαριστώ λοιπόν πρόεδρε και εγώ ίδια θα ήθελα να υπογραμμίσω εδώ το γεγονός ότι πρέπει να συναγάγουμε τα συμπεράσματά μας και τα μαθήματά μας από τα λάθη του παρελθόντος σε σχέση και με τα όσα έχουμε δει για την υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών. Έχουν υπάρξει φαινόμενα όπως επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων σε διεφθαρμένα ελιτίστικα καθεστώτα στις αναπτυσσόμενες χώρες και δεν πήγαιναν αυτά τα κονδύλια σε εκείνου που τα χρειαζόντουσαν περισσότερο, για παράδειγμα γυναίκες και άλλους θα ήθελα να παρακολουθήσουμε του σύνεγγυ, να καταστήσουμε απόλυτα σαφέ πώ μπορούμε να έχουμε μια πιο συστηματική φύση στον χαρακτήρα, συστημική φύση παρακολούθηση ε, και πώ μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι ένα σαφέ ε, σύστημα ε, δικτών θα μα κάνει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όχι μόνο να επιδοτούμε τα καθεστώτα των ελίτ, αυτό δεν σημαίνει ότι όλε οι ελίτ είναι κακές, αλλά θέλουμε να έχουμε μια ευρύτερη προσέγγιση ώστε η βοήθεια που παρέχουμε να είναι πιο αποτελεσματική και να φέρνει περισσότερα αποτελέσματα. Και γι' αυτό θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες. Και ίσως ένα τελευταίο πολιτικής υφής σχόλιο. Είναι αναγκασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεξετάσει τις πολιτικές της έναντι αυταρχικών καθεστώτων, βλέποντας τι συμβαίνει στην Λιβύη, στην Τινησία, στην Αίγυπτο. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει να δούμε τις πολιτικές επιπτώσεις που θα έχει η δράση μας και πώς πρέπει αυτή να σχεδιάζεται. Σας ευχαριστώ. Κύριος Πόρτας θέλει να προσθέσει κάτι. Παρακαλώ. Θα ήθελα να πω ότι προσυπογράφω απόλυτα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν και από την συνάδελφο ή αλλά και τη συνάδελφο Helga Τρούπερ και δεν έχω να προσθέσω τίποτα λοιπόν από αυτόν. Απλά θα ήθελα να υπογραμμίσω μια πτυχή που αναφέρεται στην ελαστικότητα, στην ευελιξία της απάντησης ε, σε σχέση με τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντί τρίτων χωρών και των πολιτικών μας. Για να δώσω ένα παράδειγμα για ποιο πράγμα κάνω λόγο συγκεκριμένα. Τώρα στην Αίγυπτο, για παράδειγμα, αυτή την ακριβή στιγμή, τώρα, σήμερα, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων, συνεχίζει να δίνει πώς να το πω εσύ να χρηματοδοτεί μη κυβερνητικέ οργανώσεις στην Αίγυπτο, που είναι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις του παλαιού καθεστώτος, του Μουμπάρακ, και εκείνες που βρίσκονται υπό την ηγεσία της συζύγου του κυρίου Μουμπάρακ. Και αυτό σε σχέση με τον πολλαπλασιασμό νέων μη κυβερνητικών οργανώσεων που βλέπουμε ότι σε παράνομο ας το πω έτσι καθεστώς συνεχίζουν να δρούν και δεν, ε, τις, ε, δεν μπορούμε να τις συνδράμουμε με κανένα τρόπο διότι είναι ιδιαίτερα α, χρονοβόρες οι διαδικασίες που υιοθετούμε και η γραφειοκρατική επιβάρηση. Ευχαριστώ. Oui, merci, cher σας ευχαριστούμε αγαπητέ φίλε όπως το επισημάνατε αρκετοί μεταξύ από εσά, νομίζω ότι πρέπει σαφώ να λάβουμε υπόψη τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρες, τον γειτονικές της Ευρώπης, ιδίως στην νότια ακτή της Μεσογείου και να κάνουμε ένα απολογισμό του τι βοήθειες δώσαμε σε χώρες όπου η κυβέρνηση δεν ήταν δημοκρατική. Ε, ως επιτοπλίστων σε αναπτυσσόμενες χώρες μάλιστα. Διαπιστώνουμε ότι συμβαίνουν τα εξής δύο τεινά είτε στην πράξη αρχές ε, εμέσως ή άμεσα φροντίζουν να πάρουν την βοήθεια στα χέρια τους, άρα έχουμε να κάνουμε δικτατορικά καθεστώτα, ή καταφέρνουμε να δώσουμε τα χρήματα τελικά στον ίδιο τον λαό, αλλά έτσι τους κάνουμε να αντέχουν ε, στα δικτατορικά καθεστώτα. Θα πρέπει λοιπόν με την ευκαιρία της έκθεσης αυτής να κάνουμε ένα συνολικό απολογισμό της πολιτικής μας και ενδεχομένως να προτείνουμε και νέους προσανατολισμούς. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την έκθεση της Αν Γένσεν, ευχαριστώ τον ε, κύριο Άγγλιν που παρουσίασε τα βασικά στοιχεία. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 15 Μαρτίου το μεσημέρι. Την δική μας ψηφοφορία θα την κάνουμε στις 31 Μαρτίου και το χρονοδιάγραμμα προβλέπει να περάσει το θέμα στην Ολομέλεια τον Ιούνιο. Εν τω μεταξύ, έφτασε ο κύριος Πέτερινγκ. Τον χαιρετίζω και τον ευχαριστώ για την παρουσία του. Το σημείο του ωστόσο προβλέπεται στις 10.30. Μας μένει ένα τέταρτο, κύριε Χάγκλουντ προλαβαίνετε σε ένα τέταρτο ως εισηγητής να μας παρουσιάσετε το σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης. Ενδιάμεσα αναθεώρηση του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα. Μπορείτε να είστε σύντομος, διότι έτσι θα καταφέρουμε να σεβαστούμε και τις πιστώσεις χρόνου που έχουμε αναλάβει. Και στις 10.30 θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Πέτρινγκ, όπως προβλέπετε. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι ο αποτελεσματικό Φινλανδό και να είμαι σύντομο. Κάνουμε λόγο για μια γνωμοδότηση λοιπόν εδώ για την αξιολόγηση αυτή τη δράση και μια και επικεντρωνόμαστε στα δημοσιονομικά μπορούμε νομίζω να είμαστε ταχεί. Έχουμε μια γνωμοδότηση που είναι σύντομη λόγω του περιορισμένου εύρου των όσων μπορούν να χρησιμοποιηθούν εδώ. Είναι πολύ σημαντικό όμω θέμα και συσχετίζεται με τα θέματα που μα παρουσίασε η συνάδελφο όσον αφορά και την έκθεση για το επόμενο έτο. Πόσο μπορούν να ευθυγραμμιστούν οι πολιτικέ μα ε, και σε σχέση με τι στρατηγικέ τη Ευρώπη 2020. Σημαντικό στοιχείο αυτό. Πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει και αυτό φυσικά θα πρέπει να είναι η αρμοδιότητα των αρμόδιων υπεύθυνων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Αλλά έχουμε και εμεί σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε εδώ. Εδώ θέλω να ξεκινήσω ω αφετηρία. Θέλω να υπογραμμίσω σε αυτή τη γνωμοδότηση ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα ευθυγραμμίζεται αυτή η πρόπτικη με τη στρατηγική του 2000, της Ευρώπης του 2020 και τι μπορούμε να συναγάγουμε από τα όσα έγιναν στο παρελθόν σε σχέση με το πολιετές αυτό πρόγραμμα. Και με τις προοπτικές για το μέλλον και να, πάρουμε, να συναγάγουμε μαθήματα από το προηγούμενο έβδομο αυτό ε, πλαίσιο και να δούμε τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Αυτό πρέπει να υπογραμμίσουμε με κάθε τρόπο. Επίσης υπογραμμίζω το γεγονός ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση ταυτοποιεί, εντοπίζει αρκετές ελλείψεις ε, όταν ε, πρόκειται για την υλοποίηση και εφαρμογή του τρέχοντος προγράμματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει ιδιαίτερα σοβαρά αυτές τις ε, παρατηρήσεις. Αυτό πρέπει να τονίσουμε με κάθε τρόπο. Πρέπει να υπάρξει η υλοποίηση με ό,τι όπως περνάει από το χέρι μας ώστε οι στόχοι να επιτευχθούν σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω την, τον επιμερισμό αρμοδιοτήτων ε, ε, για την διαχείριση προ όφελο όλων. Θα έπρεπε να υπάρχει μια βελτιωμένη πρόσβαση προ πελασιμότητα σε αυτό το μέσο, διότι βλέπουμε ότι σε κάποιε χώρες δεν είναι διαθέσιμο για την ε, έρευνα και την ανάπτυξη και όσον αφορά και τη χρηματοδότηση ένα άλλο που θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε είναι η δυνατότητα ακόμα περισσότερο να εντάσσονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ, στις πολιτικές αυτές με ένα θετικό τρόπο για να δημιουργηθεί η προοπτική της, των θέσεων απασχόλησης που θα προκύψουν και της ανάπτυξης. Επίσης λαμβάνοντας υπόψη τις υποδομές ε, για την έρευνα θα έπρεπε να διασφαλίσουμε και να δούμε πώς όλα αυτά μπορούν ε, να αποβούν προς όφελος ε, των ιδιωτικών προγραμμάτων και σχεδίων για την έρευνα. Ένα άλλο θέμα που θέλω να τονίσω είναι το γεγονός ότι ίσως είμαστε ιδιαίτερα κάπως επιφυλακτικοί με την πολιτική μας ε, για την έρευνα. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα κονδύλια για την έρευνα υψηλού κινδυνού πράγματα που μπορούν να ε, δώσουν αποτελέσματα. Ίσως εδώ είμαστε κάπως διστακτικοί, επιφυλακτικοί. Ξέρουμε ότι η έρευνα δεν δίνει πάντα αποτελέσματα, αλλά όταν υπάρχουν αυτά, αυτά είναι πολύ θετικά. Να τα λάβουμε λοιπόν υπόψη αυτά. Αυτή είναι η φύση της νομοδότησης ε, γενικά. Και θα έλεγα πρόεδρε, αυτά είναι όσα είχα να πω και επαρκούμε σε αυτά. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων στη συνέχεια για αυτό το σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Δύο ομιλητέ έχουν ζητήσει το λόγο. Θα παρακαλέσω να είστε σύντομοι. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρω ότι θέλετε να προχωρήσετε γρήγορα. Θα είμαι λοιπόν πολύ σύντομο. Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα τον κύριο Άγγλον για την έκθεσή του και τι προτάσει που έκανε. Απλώ λίγε παρατηρήσει. Πρώτον, εδώ μιλάμε για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο τη έρευνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω έχει ξεκινήσει τι διαβολεύσει για το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε απολογισμό και τα διδάγματα που θα αντλήσουμε από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο να τα χρησιμοποιήσουμε για τον προγραμματισμό του 8ου. Έπειτα, για κάποιες για κάποια ιδρύματα που ωφελήθηκαν από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο στην Ουαλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, από εκείνε τι διαδικασίε φάνηκε ανάγκη απλούστευση. Αυτό φαίνεται εύκολα και από τη συγκεκριμένη έκθεση. Πρέπει οι όλε οι διαδικασίε να απλοποιηθούν για όλου του δικαιούχου. Αλλά και κάτι άλλο που μα απασχολεί στην διαδικασία είναι εκεί που αναφέρεται η περίοδο ε, τη υποβολή αιτήσεων. Εκεί είναι πολύ σύντομη δεν υπάρχει χρόνος για την κατάρτιση των ε, κατάλληλων υποψηφιωτήτων, ούτε να αναζητηθούν εταίροι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δείτε λοιπόν περισσότερο χρόνο στα Ιδρύματα, ώστε να μπορούν να ετοιμάζουν και διασυνοριακές συνεργασίες και προγράμματα. Και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την βιομηχανία. Θέλουμε εδώ έρευνα και ανάπτυξη αλλά θα πρέπει όλες αυτές ε, οι προσπάθειες να μεταφράζονται σε προϊόντα και θέσεις εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να εμπλέξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι τα ωφέλη στο τέλος περιλαμβάνουν σίγουρα και την παραγωγή προϊόντων και θέσεων εργασίας. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστούμε. James. Ευχαριστώ. Νομίζω... Με συγχωρείτε που δεν άκουσα από την αρχή τον κύριο Χάγκλουντ στην παρουσίαση του θέματος αυτού, αλλά στην παράγραφο 6 νομίζω μιλά για απλούστευση Έχουμε ξανασυζητήσει στην Επιτροπή αυτό, τι γίνεται με τους ιστοτόπους και τους ερευνητές που δεν ε, δέχονται να συνεργαστούν στα επόμενα στάδια μιας διαδικασίας, διότι δεν έχει λειτουργήσει σωστά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας. Αυτό μας το είπε και η έκθεση του κ. Καβάλιο για την ε, ανάγκη απλούστευσης προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικές οι διαδικασίες. Εδώ πρέπει να επιταχύνουμε και τη διαδικασία επίλυσης εκκρεμουσών διαφορών. Έχουμε χιλιάδε ερευνητέ που δεν θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πλαίσιο. Κάτι, πρόγραμμα πλαίσιο. Κάτι δεν πάει λοιπόν καλά. Πρέπει να απλοποιήσουμε τι διαδικασίε αυτέ, ώστε όλα αυτά να λειτουργήσουν καλύτερα στα επόμενα στάδια του 8ου προγράμματο πλαισίου. Ευχαριστούμε, Τζέιμ. Να προσθέσω κι εγώ. Όπω είπε και ο εισηγητή, ότι το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Προκειμένου να πετύχει η στρατηγική τη Ευρώπη το 2020 για την προετοιμασία του πλαισίου του ερχόμενου προγράμματος για όλου αυτού του λόγου πρέπει να κάνουμε έναν καλό απολογισμό του πώ λειτουργεί το τρέχον πρόγραμμα. Ήθελα λοιπόν εδώ να δώσω τη δική μου μαρτυρία και ίσω και να αποβάλω και σχετική τροπολογία. Να πω το εξή. Στην περίπτωση τη Γαλλία, ένα πολύ μικρό μέρο των ερευνητικών προγραμμάτων ευρωπαϊκής διάστασης αφορούν ε, ιδιωτικά ή κρατικά ερευνητικά κέντρα της Γαλλίας. Γαλλία. Κειμιλήσει σχετικά καλά το σύστημα. Έχουμε όμω και εθνικό που είναι 4 ή 5 φορές ε, υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Κάτι που ισχύει για πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Διαπιστώνω λοιπόν ότι η χρήση, του προπολογισμού στη Γαλλία για ερευνητικού σκοπού δείχνει τάσει ε, να είναι παροχημένο ω προ τη δικασία. Ε, δεν συζητούν οι φορεί δημόσιοι και ιδιωτικοί. Όλε οι προσπάθειε λοιπόν που είναι επικοδομητικέ ε, από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Προγράμματο Πλαισίου και έχουν γίνει ώστε τα ερευνητικά κέντρα να συνεργάζονται μεταξύ του, δεν εφαρμόζονται σε όλου του ερευνητέ μα. Και αυτό το, πρόγραμμα, το πνεύμα που προσπαθήσαμε να εμφυσίσουμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο δείχνει ότι πρέπει να διορθώσουμε σφάλματα, να καλύψουμε κενά, αλλά τώρα πρέπει να το εμφυσίσουμε και στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων μας, που είναι αποκλειστικά εθνικού χαρακτήρα. Αυτό ήταν το πνεύμα της έκθεσης και της κυρίας Μπαλτιάνη βρίσκεται και στο κέντρο των μεριμνών της Επιτροπής Σούρα. Πρέπει να δούμε πώς θα αξιοποιούμε καταλήλως στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και πώς θα δίνουμε από κοινοτική πλευράς το παράδειγμα στα εθνικά κράτη-μέλη, ώστε να εμπνέονται και να μπορούν να συνεργάζονται σε ένα διακυβερνητικό πλαίσιο. Και στην δική τους τη διαχείριση να αντλούν τα, και να αξιοποιούν τα μαθήματα που έχουν αντλήσει από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Κυρία Σιτά, θέλετε να κάνετε κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, συνάδελφοι, για τα σχόλια. Επιτρέψτε μου να πω ότι θα υπάρξει και μια πρόσθετη γνωμοδοσία για το πρόγραμμα πλαίσιο, το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο που θα ακολουθήσει. Και έτσι θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό υστερότερα, σχετικά σύντομα. Ευχαριστώ. Très bien, merci. Donc, je... Ευχαριστούμε. Θυμίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ορίζεται στι 16 Μαρτίου στι 4. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Προπολογισμών την έκθεση στι 31 Μαρτίου. Η Επιτροπή Ήτρε, που είναι υπεύθυνη επί τη ουσία, θα ψηφίσει κατά πάσα πιθανότητα στη συνεδρίαση τη 12η-13η Απριλίου. Προκειμένου η ψηφοφορία στην Ολομέλεια, που είναι προ επιβεβαίωση, να γίνει τον Μάιο. Φτάνουμε λοιπόν εγκαίρως στο σημείο 6, ακριβώς τη στιγμή που προβλεπόταν. Ανταλλαγή απόψεων με τον Αντιπρόεδρο Μαρτίνες Μαρτίνες, τον οποίο χαιρετώ, και τον Πρόεδρο κ. Χάνς Γκέρτ Πέτερινγκ. Χαίρομαι πολύ που τον ξαναβλέπω. Να πω στους συναδέλφους ότι είχαμε την τιμή πριν λίγες εβδομάδες στο μέγαρο του Ελιζέ των Λυσίων στο Παρίσι να φιλοξενήσουμε τον κύριο Πέτερινγκ και έλαβε το παράσημο της Λεγιώνας ε, στο Παρίσι. Ε, και αυτό είναι ένα ορόσημο για τη συνεργασία Γαλλίας και Γερμανίας. Χαιρετίζω λοιπόν όλα τα μέλη της ομάδας αυτής που δίνουν ζωή στο όλο σχέδιο για τη δημιουργία του, του σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Έχει παρουσιαστεί το σχετικό σχέδιο στα μέλη της Επιτροπής. Η κυρία Τρίπελ θα ήθελε το λόγο σε αυτό το στάδιο ή να ακούσουμε τους συντάκτες του σχεδίου να μας το παρουσιάζουν και μετά να κάνετε τα σχόλιά σας. Προφανώ οι συνάδελφοι που θέλουν θα μπορούν να θέσουν και ερωτήσει. Εδώ έχω μια υπέροχη φωτογραφία. Την έχετε δει όλοι. Α, μόλι τη μοιράζουν. Δεν έχουμε δυστυχώ βίντεο wall. Δεν ξέρω ποιος θα πάρει το λόγο. Ο Χανσκέτη ίσω. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Αλέλα Μασούρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι πραγματικά χαρά να μπορώ να παρίσταμαι εδώ. Τον Ιούλιο 32 μέλη θα είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1979 από τις πρώτες άμεσες εκλογές. Ποτέ δεν είχα τη χαρά και κυρίως δεν είχα την τιμή σε αυτή την πολύ σημαντική Κοινοβουλευτική Επιτροπή να λάβω τον λόγο και να σας προσφωνήσω. Σήμερα είναι η πρώτη φορά αυτή και μια και αυτό είναι η πρώτη φορά είναι μια, ένα ιδιαίτερο βίωμα, μια ιδιαίτερη εμπειρία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά λοιπόν για τα συγχαρητήρια του Προέδρου σας, του Αλέλα Μασού του Αλέν Λαμασούρ για αυτό το γεγονός στο μέγαρο των ηλισίων. Επιτρέψτε μου να προσθέσω, όταν προσήλθα στην αίθουσα γινόταν λόγος για τις αραβικές χώρες. Αύριο θα πάω υπό άλλη διαφορετική ιδιότητα για τρεις μέρες στην Αίγυπτο, στο Κάιρο, ώστε το δημοκρατικό κίνημα να το υποστηρίξω εκεί. Γιατί το λέω αυτό. Το λέω επειδή για το θέμα αυτό κάνει μια καλή εισαγωγή μας εισα... μπορεί να μας ε, ε, εισαγάγει στο θέμα αυτό με καλό τρόπο, το θέμα το οποίο συζητούμε, τον οίκο της ευρωπαϊκής ιστορίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, συζητάμε πολλές φορές, πολύ συχνά, μόνο για οικονομία, χρηματοοικονομικά θέματα και στην Ευρώπη. Και έχω την εντύπωση ότι για το ουσιώδες, για το οποίο συνενωνόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χάνουμε ενώπιόν μας αυτό το σημαντικότερο στόχο. Είμαστε συνενωμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 550 εκατομμύρια πολιτών με βάση κοινέ αξίες και αρχές και ακριβώ αυτό πολύ λίγο το συνειδητοποιούν οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ω στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται μόνο για κονδύλια, χρήματα, ε, οικονομικά, χρηματοοικονομικά θέματα και γεωργία, όσο σημαντικά και αν είναι αυτά, αλλά για τι κοινέ αξίε και αρχέ που μα συνενώνουν. Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, δυνατότητα δημοκρατική διαβίωση. Και θέλουμε με έναν οίκο τη Ευρωπαϊκή Ιστορία να πετύχουμε ακριβώ αυτό το στόχο. Για του πολίτε μα, κυρίω για του νέου μα πολίτε, να καταστήσουμε σαφή αυτή τη διάσταση. Και γι' αυτό πρότεινα τον ε, Φεβρουάριο ήδη 2007 στον προγραμματικό μου λόγο ως Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τότε ότι ένα τέτοιο οίκο της ευρωπαϊκής ιστορίας θα έπρεπε να δημιουργούσαμε, είχα πει. Και αυτό έχει και επιστημονικό συμβούλιο το οποίο παρακολούθησε Συμβούλιο Πραγματογνωμόνων Επαϊόντων για το σχέδιο που υπέβαλαν στη συνέχεια για τη δημιουργία αυτού του οίκου Ευρωπαϊκή Ιστορία. Όλα αυτά τα στοιχεία τα έχετε στη διάθεσή σα. Και θα ήθελα να πω ότι ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα και χαίρομαι για το ότι ο Αντιπρόεδρο ε, Μιγέλ Άγχελ Μαρτίνεθ Μαρτίνεθ είναι παρόν και συνεργαζόμαστε και εργάζεται και αυτό από κοινού για αυτό το εγχείρημα, από κοινού με άλλου όπω και εγώ. Υπήρξε μια τέτοια λοιπόν συνδρομή Συμβουλίου Επαϊόντων και τις γνώσεις του ή τις, ε, τα συμπεράσματά του τα συνεπέρανε σε μια πρόταση που λέει ότι θέλουμε τις γνώσεις των Ευρωπαίων να τις διασφαλίσουμε για όλες τις γενναίες, για την ιστορία και να εμβαθύνουμε σε αυτή την ιστορία ώστε να συνεισφέρουμε σε αυτή τη χρονική στιγμή εμείς προς αυτή την κατεύθυνση. Ο οίκος της ευρωπαϊκής ιστορίας θα έχει ως κύριο βάρος, κύριο βάρος την ιστορία του 20ου αιώνα με τις τραγωδίες, τα ολοκληρωτικά συστήματα εξουσίας, τους παγκόσμιους πολέμους και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει πολλαπλά να αναφερόμαστε στην ευρωπαϊκή ιστορία και πριν από τον 20ο αιώνα αλλά και σε αυτόν. Δημιουργήσαμε συντονιστές και κοσμήτορες. Αυτά ήταν αποφάσεις ε, του ε, Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εννέα φορές ασχολήθηκε το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια ομάδα κοσμητόρων υπό την δική μου ηγεσία και του αναπληρωτή ε, Προέδρου Μιγελ Άγχελ Μαρτίνεθ Μαρτίνεθ όπου όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντανακλώνται και με τον Ζεράρο η με τον Ευρωπαϊκή Συντηρητική και Μεταρρυθμιστέ, με την Αντιπρόεδρο κυρία Νταϊάννα Γόλης η Φιλελεύθερη, η ε, Αριστερή επίσης και με τον Αλέν Λαμασούρο Πρόεδρο τη Επιτροπής Προϋπολογισμών που ανήκει σε αυτό το όργανο και εκείνο έχουμε ένα επιστημονικό συμβούλιο υπό την Προεδρία ενός ε, ε, Πολωνού ιστορικού του Σίμιετς Ροσδέη ενός αναγνωρισμένου ιστορικού και έχουμε και πολλούς άλλους ε, επαΐοντες ε, άξιους ιστορικούς ε, που συμμετέχουν. Θέλουμε διαφάνεια. Θέλουμε να προχωρήσουμε με αυτό το πλαίσιο όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Μην αναμένετε όμως απαντήσεις αγαπητοί συνάδελφοι που δεν μπορούμε να δώσουμε σήμερα όσον αφορά και το 2018 ή 2020. Θέλουμε μέχρι τότε να μπορέσουμε να απαντήσουμε όσο το καλύτερο γίνεται και αποφύγαμε και στην δημοσιότητα τέτοιου είδους ε, πρωτοβουλίες ε, διότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε, να ακολουθήσουμε τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ο πρόεδρος Μπούσεκ προτείνει για το Προεδρείο το αποθεματικό των 2,5 εκατομμυρίων που χρειαζόμαστε για την προσυπογραφή του, ε, της συμφωνίας με τους αρχιτέκτονες να απελευθερωθεί αυτό το κονδύλιο και αυτή είναι η παράκλησή μας προς εμάς να συνδράμεται να απελευθερωθεί αυτό το κονδύλιο. Έχουμε και 26 αρχιτέκτονες που συμμετείχαν στην αρχική προκήρυξη. 12 στη συνέχεια επελέγησαν από μια διαδικασία πρώτη επιλογή για προτάσει του. Στο τέλο, δύο απέμειναν στην τελική επιλογή. Και είχαμε πρόσφατα, ε, προχθέ το βράδυ, μία ε, σύγκληση υπαλλήλων που έλαβαν την τελική απόφαση για ένα γραφείο αρχιτεκτόνων Τζένι Μορέλ είναι ένα γραφείο αρχιτεκτόνων που και το πτή παλέ, το μικρό μέγαρο στο Παρίσι, το είχαν ε, μετασκευάσει. Είχαμε και μια μικρή ομάδα συνεργατών, γυναικών και ανδρών, που ασχολήθηκαν με το πρόγραμμα αυτό επιστημονικά και η διευθύντρια, κυρία Ιτάλια και Φανγκάλ, είναι η κυρία εδώ, που δεν είναι απόλυτα στα κόκκινα ενδεδειμένη αλλά με βάση το χρώμα αυτό ε, των, ε, ε, της αμφίεσής της θέλω να την επισημάνω είναι η διευθύντρια, είναι ε, σλοβενικής υπηκότητας και συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα εργασιών. Τώρα αγαπητοί συνάδελφοι για αυτά τα οποία θεμητά εσείς έχετε ως αρμόδιοι για τα δημοσιονομικά θέματα ιδιαίτερα υπόψη σας το κόστος δηλαδή αυτά τα οποία εσείς εξετάζετε εργαστήκαμε με βάση υγιή κριτήρια και 31 εκατομμύρια ευρώ θα χρειαστούν για την ε, μετασκευή και της, ε, την ανακαίνιση και την διεύρυνση του επέκταση του κτηρίου Eastman. Σημαντικό αυτό, επέκταση του κτηρίου Eastman. Γνωρίζετε το κτίριο Eastman στο Πάρκο Λεοπόλδου. Υπάρχει ένας ε, ελεύθερος χώρος πίσω από το κτίριο και θα πρέπει εκεί να υπάρξει επέκταση όταν θα υπάρχει η αναγκαία προηγούμενα απόφαση. Έχετε και τα σκαρίφημα, τα σχέδια που σας έχουν διατεθεί μετά θα χρειαστούμε 21,4 εκατομμύρια ευρώ για την διαμόρφωση της ε, ε, διαρκούς έκθεσης και της έκθεσης στους χώρους ε, των κτηρίων αυτών, ώστε 21,4 εκατομμύρια ευρώ να χρειαστούν για την εσωτερική ας το μουσιακά αυτού του κτηρίου. 3 εκατομμύρια επιπλέον θα χρειαστούν στη συνέχεια για τη συλλογή και την ε, παρουσίαση των αντικειμένων που μέσα σε, αυτό, αυτή την έκθεση θα παρουσιαστούν. Υπάρχουν εκτιμήσεις δαπανών επίσης για την ε, διαρκή λειτουργία. 6 7 εκατομμύρια για μόνιμα έξοδα ε, ε, θα έχουμε και την μόνιμη έκθεση, της επιμέρους εκθέσεις την, τον καθαρισμό, την θέρμανση, τα θέματα διαρρύθμιση δεν έχουμε λάβει υπόψη τι γενικέ ε, υπηρεσίε, ε, τα σημεία ενημέρωση και τέτοιου είδου λεπτομέρειε. Αλλά σε στενή συνεργασία με τι ε, ήδη υπάρχουσε υπηρεσίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εκτιμηθούν και θα σα παρουσιαστούν. Θα έχουμε λοιπόν ανάγκη 18 στελεχών όσον αφορά τη διοίκηση και 18 βοηθών σε σχέση με τις εργασίες που πρέπει να καλυφθούν. Πρόκειται για υπαλλήλου με συμβάσει προσωρινής απασχόλησης, προσωρινού χαρακτήρα. Είναι αυτονόητο ότι όλα αυτά θα είναι διαθέσιμα όταν θα έχει ληφθεί, όταν θα ληφθεί πρώτα η θεμελιώδης απόφαση απελευθέρωσης του κονδυλίου και σε σχέση και με το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με ερώτηση που έκανα μου το επιβεβαίωσαν. Όλα αυτά μέσα από την έννοια της γνωστοποίησης ή ενημέρωση. Δεν γνωρίζω ποια είναι η σωστή ορολογία, αλλά μέσα από τις τυπικές και επίσημες διαδικασίες ε, γραπτά και όπως προβλέπετε θα διαβιβαστούν αυτά τα στοιχεία προς έγκριση. Ο οίκος ευρωπαϊκής ιστορίας πολυσχηδεί μέσα για την επικοινωνία θα χρησιμοποιεί. Θα έχουμε έκθεση πολυμέσων, προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και επιμόρφωσης ώστε να δίνεται μια προοπτική της ιστορίας ε, σε αυτές τις δράσεις. Θα έχουμε και εμβαδόν 4.000 τετραγωνικών μέτρων και θα έχουμε και μια περιφερόμενη προσωρινή έκθεση σε 800 τετραγωνικά μέτρα. Έτσι θα μπορεί να δημιουργηθεί ένα δίκτυο, μουσιακό δίκτυο με εθνικά μουσεία στις χώρες μέλη, ώστε έτσι η προοπτική της Ευρώπης στο ιστορικό επίπεδο, στο εθνικό όμως επίπεδο των κρατών μελών, να μπορεί να συμπληρώνει εκθέσεις σε μουσεία που υπάρχουν στα κράτη-μέλη, ώστε να να αντανακλάται η ευρωπαϊκή ιστορία. Έτσι λοιπόν νομίζω, μια και πρέπει να, διατηρήσω το, να τηρήσω το όριο των 10 λεπτών που προβλέφθηκε, πρέπει να πω αγαπητοί συνάδελφοι, ο οίκο ευρωπαϊκής ιστορίας είναι τμήμα μια σύγχρονη στρατηγική για επισκέπτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με άλλα λόγια, οι επισκέπτε στα θεωρία, οι επισκέπτε αυτοί για αυτούς αυτή η πτυχή θα έχουν, για αυτή την πτυχή θα έχουν το γραφείο ε, πληροφόρησης και δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ του κέντρου πληροφόρησης και του οίκου ιστορίας. Το οίκο ε, πληροφορι... Ο οίκος πληροφοριών, το κέντρο πληροφοριών θα πληροφορεί για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, για το πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ ο οίκος Ευρωπαϊκής Ιστορίας θα ασχολείται και θα καλύπτει την ιστορία και πώς καταλήξαμε στη σημερινή Ευρώπη σήμερα, στη σημερινή συγκυρία και ποια πορεία θα ακολουθήσει αφήσουμε στο μέλλον. Οι επισκέπτε προσέρχονται δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορούν να επισκέπτονται το κέντρο επισκεπτών, να έχουν και την επαφή με το κέντρο πληροφοριών, μπορούν να γνωρίζουν και να επισκέπτονται και το, ε, τον οίκο Ευρωπαϊκή Ιστορία. Όλα αυτά είναι τμήματα ενό συνολικού προγράμματο για επισκέπτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έτσι όταν έρχονται εδώ επισκέπτε, ε, ομάδε και επισκέπτονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουν τέτοιε δυνατότητε, θα χρειάζονται και ένα κηλικείο. Θα υπάρχει κηλικείο στον οίκο Ευρωπαϊκής Ιστορίας, ώστε έτσι στο ίδιο το κτίριο, περνώντας από τους διαδρόμους και επισκεπτόμενοι τους χώρους εκθέσεων, οι επισκέπτες, να μην στριμώχνονται, να μην έχουν προβλήματα, να μπορούν να επισκέπτονται την καφετέρια και να έχουμε την δυνατότητα να επισκέπτονται στη συνέχεια και τον οίκο Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Θα ήθελα να πω στη συνέχεια, όταν τίθεται το ερώτημα, τι γίνεται για τη χρηματοδότηση του οίκου Ιστορίας μέσω άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Θα ήθελα σε εσά να πω και η πολιτική είναι, αυτό είναι το βίωμά μου μετά από 32 χρόνια προπηρεσία εδώ, η πολιτική είναι θέμα εμπιστοσύνη. Αν τώρα εδώ σε αυτό το θέμα Συμβούλιο Υπουργών και Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είχαν εμπλακεί και ρωτούσαμε ποια κονδύλια θα δίνατε εσεί κύριοι, θα είχε αποτύχει αυτό το ε, εγχείρημα. Δεν θα είχαμε απαντήσει από τα άλλα θεσμικά όργανα. Γι' αυτό το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νομίζω και με την υποστήριξη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων ήταν στο, στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό ο οίκο Ευρωπαϊκή Ιστορία θα είναι το δικό μας εγχείρημα, η δική μας πρωτοβουλία. Εμείς θα το καλύψουμε, ιδιαίτερα τους νέους στους επισκέπτες και στους νέους θέλουμε να στραφούμε. Και έτσι θα είναι υπόθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτός ο οίκος Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Ως τμήμα, μέρος μιας σύγχρονης ε, πολιτικής για τους επισκέπτες ε, στο Ευρωκοινοβούλιο. Φυσικά κανείς μπορεί να προβληματιστεί. Και εγώ ίδιος προβληματίζομαι αλλά και για το Προεδρείο και εσάς ε, κύριε Μιγέλ Άγχελ Μαρτίνεθ Μαρτίνεθ και εσάς Ιζαμπέλ βλέπω που εργάζεστε σε αυτό το εγχείρημα στο Προεδρείο. Πρέπει να εξεταστεί το θέμα ποια θα είναι τα κόστη κόστη, επακόλουθα κόστη, όταν θα δημιουργηθεί ο οίκος Ευρωπαϊκής Ιστορίας ποια θα είναι τα υπακόλουθα κόστη σε σχέση με τον επιμερισμό, σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και πώς θα μπορούν να επιμεριστούν αυτά τα κόστη αναμεταξύ μας. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει και θα μας προβληματίσει για το μέλλον. Αλλά από πλευράς ε, κοσμητόρων και υπεύθυνων για αυτό το νίκο Ευρωπαϊκή Ιστορίας θέλουμε να σας πούμε ότι με απόλυτη διαφάνεια θα διεξαχθούν όλα αυτά. Θα σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες που μπορούμε να σας δώσουμε, αλλά δεν μπορούμε σε όλα τα ερωτήματα να έχουμε σήμερα τελικές ειδικές απαντήσεις. Αν υπάρχει καλή πρόθεση και προαίρεση μπορεί να προχωρήσει αυτό το εγχείρημα και να ευδοκιμήσει και για τις νέες γενναίες, μελλοντικές γενναίες θα μπορέσουμε να τις συνδράμουμε όσον αφορά την ιστορία της Ευρώπης. Γι' αυτό σας παρακαλώ το αποθεματικό το οποίο υπάρχει <clears throat> να το απελευθερώσετε για τα 2,5 εκατομμύρια να απελευθερωθούν αυτά ώστε η συμφωνία να υπογραφεί με το Γραφείο Αρχιτεκτόνων και να προχωρήσει αυτό και από κοινού να προχωρήσει προχωρήσουμε στη δημιουργία του οίκου Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο μέλλον. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή και κατανόησή σας. Σας ευχαριστώ εσάς ε, ιδιαίτερα θερμά για την προσοχή σας και όπως ελπίζω και εύχομαι για μια καλή συνεργασία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Merci beaucoup, cher Hans Gerd de cette présentation qui Σας ευχαριστούμε κύριε Hans-Gert Pöttering για αυτή την σαφέστατη παρουσίαση και για όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία μας διαθέθηκαν, διατέθηκαν εδώ στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Βλέπω ότι και ο Αντιπρόεδρος κύριος Μιγελάν Ματίνες Ματίνες θέλει να παρέμβει. Παρακαλώ συντομία στην παρέμβασή σας διότι πρέπει να προχωρήσουμε και σε ψηφοφορία. Ο κύριος Ματίνες Ματίνες. Επίσης θα ήθελα να σας πω Να σου πω κάποια πράγματα Διαφορετική ε, φύσεω και, και, και, και κάπως συμπληρωματικά να σα τα πω ή στα ισπανικά. Συνεχίζει ο κ. Μαρτίνε στα ισπανικά. Θεωρώ ότι αυτή η πρόκληση που αφορά το μουσείο είναι το ότι θα πρέπει έτσι να αναδείξουμε κάτι το οποίο όταν το λέμε αυτό τώρα, ε, όταν το λέω αυτό σε συμπατριώτε μου, θα πρέπει να, να, να σα πω ότι το παρουσιάζω σαν περίπου ένα θαύμα. Ένα θαύμα το οποίο τι πάει να πει, ότι έχουμε ένα σωρό αιώνε που περάσαμε με αυταρχικό καθεστώ και μετά μετασχηματισμό έγινε προς την δημοκρατία. Από τη δυστυχία στην ευημερία. Από την αντιπαράθεση στην ολοκλήρωση, στην ενοποίηση και από τον παραλογισμό, την τρέλα του πολέμου περάσαμε στην ε, λογική, στην υφαλιότητα της ειρήνης. Όχι, δεν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με, με, με κανένα Θεό. Είναι θέμα πολιτικής και των πολιτικών ή στην υπηρεσία των λαών τους και ελεγχόμενοι από τον λαό τους. Οπότε αυτό γίνεται τώρα και δεν είναι μία σύμπτωση ότι γίνεται σε μία τέτοια συγκυρία. Μία συγκυρία για το πώς η πολιτική και η πολιτική με όμικρον γιώτα πρέπει με κάθε ευκαιρία να αποδεικνύουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να κάνουμε τέτοια θαύματα όπως αυτό που σας προανέφερα. γιατί ένα δεύτερο πρόβλημα είναι εάν αυτό το θαύμα είναι αναστρέψιμο. Γιατί αυτό το πιστεύουν πάρα πολλοί από τους νέους που έρχονται εδώ, ξέρουν για τις Βεξέλλες. Όχι, δεν είναι ένα θαύμα αναστρέψιμο ή ανατρέψιμο ή είναι κάτι που έχει παγιωθεί, έχει στεριώσει. Και πρέπει κανείς να το καταλάβει, να το ξέρει και να το προστατεύει γιατί τίποτα δεν μας εγγυάται, δεν, μας, δεν καθιστά σίγουρο το ότι μπορεί κανείς να ξαναγυρίσει από τη λογική στον παραλογισμό. Οπότε θα πρέπει να σας πω ότι δεν είναι προσέγγιση το ότι αυτή ε, την, την, την, ε, την πρωτοβουλία δεν είναι καθόλου τυχαίο που τα έλαβε το κοινοβούλιο. Αφορά υπόθεση μιας 20 ετίας που αυτό κουβεντιαζόταν. Είναι κάτι το οποίο επί 15 ετία δεν γινότανε. Και αυτό γιατί όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει. Και πολλές φορές οι κοκόροι μαλώναν μεταξύ τους. Και επομένως ε, αποδείξαμε ότι έχουμε αντιπροσωπευτικότητα, έχουμε τη συνένεση ούτω ώστε ακριβώς να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς αυτή την υπόθεση και λέω να προχωρήσουμε γιατί ακριβώς το, το Κοινοβούλιο όσον αφορά αυτή την υπόθεση δεν έχει το ρόλο του να κάνει ε, αυτό το μουσείο ε, κομμάτι, τμήμα, παράρτημα του Κοινοβουλίου. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να ξεκινήσει αυτή η υπόθεση, αυτό το μουσείο να, να, να, να, πάρει το, δρόμο του και να ε, έχει την λειτουργία του, να έχει την, την αυτάρκειά του και σε λειτουργία και σε οικονομικά. Και αυτό επομένως είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Οπότε, και εμεί είμαστε υποχρεωμένοι αυτό το παρουσιάζουμε στον κόσμο και επίση και κάτι άλλο σκεφτείτε, ότι όταν ανοίγει ένα μουσείο, το πρώτο πρόβλημα για όλα τα μουσεία είναι το ποιοι, πόσοι θα έρθουν. Όμω εδώ δεν έχουμε πρόβλημα. Εδώ έχουμε ένα εκατομμύριο κόσμο που στα, στα εγγένεια κάνει ουρά για να μπει στο μουσείο. Τόσοι έρχονται. Τόσοι έρχονται καλεσμένοι μας. Και κάθονται και περιμένουν για να μπουν στο μουσείο από όλες τις χώρες και από χώρες άλλες που δεν είναι οι δικές μας γιατί ακριβώς θέλουμε να δείξουμε και σε χώρες που θέλουν να αποκτήσουν αυτή την ελευθερία όπως οι χώρες της Βορειοαφρικής ότι είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια φαινόμενα όπως αυτά τα οποία γνωρίσαμε εδώ στην Ευρώπη οπότε έρχονται και αυτοί και θα έρθουν για να επισκεφθούν το μουσείο γι' αυτό σας λέω ότι, ότι πρώτα πρώτα ε, οι νέοι πρόκειται να έρθουν αλλά και λιγότερο νέοι γιατί αυτό είναι κομμάτι της ζωής μας. Πολλοί λοιπόν θα έρθουν και για να δούνε πώς ξεκίνησαν όλα αυτά. Εκεί που λέει η ζωή μου ποτέ πια δεν ξεχνώ και λοιπά. Πρόκειται για αυτή τη ε, διαδικασία της ε, συμφιλίωσης, της προσέγγισης. Πρώτα πρώτα Γάλλη και Γερμανία. Όπως επίσης και μια σειρά των χωρών της Δυτικής Ευρώπης που έχουν περάσει από κυβερνήσεις φασιστικές γιατί δεν ήταν δυνατόν ούτε οι Πορτογάλοι, ούτε οι Έλληνες, ούτε οι Ισπανοί να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε αυτή τη διαδικασία που εσείς είχατε το προνόμιο να την κάνετε, να την περάσετε. Άλλοι για τον ένα λόγο, άλλοι για τον άλλο, ε, άλλοι γιατί είχαν δώσει τη μάχη τους στην αντίσταση, οπότε έτσι θα καταδειχθεί πως η Ευρώπη, η Δυτική και η Ανατολική έδωσε τη μάχη της τόσο ώστε να ξεπεράσει την, ε, τον αυταρχισμό ολοκληρωτικά καθεστώτα της δικτατορίας και επομένως ε, έτσι θα υπάρξει ταύτιση με το ευρωπαϊκό όραμα και θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η υπόθεση του μουσείου, του μουσείου να μην θεωρηθεί ένα κάτι, κάτι περιττό, ένα διακοσμητικό στοιχείο είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης είναι σημαντικό το, να έχουμε και τη συμπαράσταση όλων των ε, μελών, των συναδέλφων της Επιτροπής των Προϋπολογισμών και να μην κολλάμε σε λεπτομέρειες. Το είπε ο κύριος Πέτερινγκ βεβαίως, ότι όλες οι πληροφορίες, οι απαραίτητες είναι στη διάθεσή σας και δεν θέλουμε να κάτσουμε να, να, να, βυζαντινολογήσουμε για θέματα τα οποία δεν, δε λύνονται, ερωτήσεις χωρίς απάντηση. Αυτό επομένως και τέτοιο, αυτή η όθηση να δοθεί στα πράγματα Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε, λέει ο πρόεδρο τη Επιτροπή. Και τώρα, Ελγα, έχει ζητήσει το λόγο τώρα ή θε πρώτα να ακούσει συναδέλφου. Να ακούσουμε του συναδέλφου, ναι. Ποιο θέλει το λόγο. Α, θέλει το λόγο τώρα. Α, συγγνώμη, συμπάθαμε. Χέλγα. Η κυρία Τρούπερ, ναι, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πέτερν και εσάς κύριε Μαρτίνεθ Μαρτίνεθ για τις επεξηγήσεις σας. Θα ήθελα να σας πω ξεκάθαρα και να το πω επίσης και προς τους άλλους ευρωβουλευτές συναδέλφους ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού από την ιδέα και προσέγγιση αυτού του σώματος ε, δεν είχα πιστεί Πιστεύω ότι αυτή η προσέγγιση να δημιουργηθεί ένα οίκο ευρωπαϊκή ιστορία με όλα τα επιχειρήματα που εσεί εκφράσατε το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό, αναγκαίο και πάρα πολύ ευκταίο και ο τρόπος με τον οποίο το Επιστημονικό Συμβούλιο δημιουργήθηκε και συστάθηκε και με τέτοια πολυσχηδή ε, σύνθεση δημιουργήθηκε είναι σημαντική συνεισφορά. Και επίσης και η ιδέα με το διαδίκτυο, τη δικτύωση με μουσεία σε, άλλους, ε, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ανατολική Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ευρώπη, να συνεισφέρουμε για την πολυμορφία της ιστορίας στην ε, Ευρώπη ε, είναι πάρα πολύ θετικά. Επαρκούμε σε αυτά. Τώρα, για να σας πω τους άλλους λόγους τώρα, γιατί τους λόγους της Επιτροπής Προϋπολογισμού και μια και μιλάμε για προϋπολογισμού, να το πω ξεκάθαρα. Έχουμε συνολική ευθύνη εμείς όσον αφορά τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου και πέρσι για τον προϋπολογισμό του 2011, τον δικό μου προϋπολογισμό 2011 για το Ευρωκοινοβούλιο, είχα πει ότι κάποιες αυξήσεις είναι απόλυτα αναγκαίες για τις συνθήκες Λισαβόνας, αλλά σε περίοδο συγκυρία κρίσης πρέπει να δείξουμε στους πολίτες μας ότι είμαστε πρόθυμοι για αυτοπεριορισμούς και αυτοπιθαρχία, διότι διαφορετικά παρακολύεται η, αποδεκτικο... η αποδοχή από τους πολίτες. Ο κύριος ε, Φερνάντεθ για τον προϋπολογισμό 2012 έθεσε την προοπτική παγίωσης ε, του προϋπολογισμού. Παγίωση. Να το πάρουμε σοβαρά αυτό. Αν θέλουμε να παγιώσουμε και να εξηγιάνουμε, πρέπει να υποβάλουμε προτάσεις πού θα παγιώσουμε. Και δεν μπορούμε να έχουμε πάσης φύσεως προτάσεις όπου περισσότερες δαπάνες θα προκληθούν. Με άλλα λόγια, αν εμεί θέλουμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ω Επιτροπή Προπολογισμών ότι συνιστούμε την ε, υλοποίηση αυτού του προγράμματο, πρέπει πιστεύω να υπάρξουν περικοπέ σε άλλα σημεία, ώστε ο στόχο τη υπευθυνότητα, τη παγίωση του προπολογισμού και τη αυτοπιθαρχία να υλοποιηθεί. Στη σημερινή συγκυρία αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο. Επίσης θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο, ότι για την πολιτική κτηρίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπήρξε πίεση να υπάρξει μεσοπρόθεσμα σχεδιασμό κτηριακή πολιτικής. Το ίδιο κριτήριο πρέπει να ισχύει και για μας ως Ευρωκοινοβούλιο όμως και απόλυτα με διαφάνεια και υπευθυνότητα να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα νέων κτηρίων που θέλουμε να δημιουργήσουμε και πώ χρηματοοικονομικά θα καλύψουμε όλες αυτές τις ανάγκες. Δεν μπορώ να κατανοήσω απόλυτα το γεγονός ότι εμείς πρέπει ως Κοινοβούλιο εμείς αποκλειστικά μόνοι μας να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία του οίκου ευρωπαϊκής ιστορίας όπου, μια και είναι ένα βαθύτατα ευρωπαϊκό εγχείρημα και πρέπει να υποθέσουμε και να πούμε ότι και, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο θα, υπάρχει, πρέπει να υπάρχει συμμετοχή μια και εκείνοι πρέπει να αποδεχθούν την ε, σημασία, τη σπουδαιότητα αυτού του εγχειρήματο. Πώς μπορεί διαφορετικά να αντιμετωπιστεί ένα θέμα παρά διοργανικά για ένα τέτοιο εγχείρημα. Δεν μπορούμε εμεί μόνοι μα να το αναλάβουμε. Έχω και κάποια θέματα λεπτομέρεια στη συνέχεια που θέλω να αντιμετωπιστούν και θα ήθελα να απο απαντηθούν. Για τα επιμελητιακά θέματα. Οι πολλοί ε, επισκέπτε που ελπίζουμε ότι θα προσέλθουν στο Ευρωκοινοβούλιο θέλω να ξέρω πού θα σταματούν τα λεωφορεία, πού θα είναι η στάση του, να μην υπάρχουν στενοποί και προβλήματα και ατέλειωτα προβλήματα. Μετά για το transfer, τη μεταφορά, για την απελευθέρωσή του, για τα 2,5 εκατομμύρια. Πού θα τα χρειαστείτε ακριβώ, για την σύμβαση που θα υπογράψετε με το Γραφείο Αρχιτεκτόνων. Αυτά που έχουμε μελέτε από τους αρχιτέκτονες μέχρι σήμερα αυτά τα σχέδια έχουν πληρωθεί ήδη ή πρέπει να πληρωθούν ακόμα. Πώς γίνεται δηλαδή η χρήση, με τις μέχρι, η πληρωμή της μέχρι σήμερα εργασίας που έχει γίνει. Ποια μορφή έχει. Θα ήθελα να απαντηθεί. Και τελευταία ερώτηση. Ποια είναι η αναλογία. Ποια είναι η αναλογία. Το αναφέρατε αλλά θέλω ε, ξεκάθαρα να το πω μεταξύ των συντονιστών και κοσμητόρων όπου είναι ο κύριος ε, Πέτερινγκ και του Επιστημονικού Συμβουλίου. Ποιος είναι ο συσχετισμός τους σε σχέση με την πολιτική κατεύθυνση που ακολουθείτε σε σχέση με αυτό το εγχείρημα. Αν μπορείτε να μας τα επεξηγήσετε σύντομα. Ευχαριστώ. Ο πρώτος, σας ευχαριστώ. Οπότε παρακαλώ οι συνάδελφοι να η πιο σύντομη όταν το λόγο. Σαλβαντόρ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η ομάδα μας δεν έχει υπερβολικά προβλήματα να δεχτεί την απελευθέρωση αυτού του αποθεματικού ποσού. Ωστόσο όμως παρόλα αυτά και εγώ συμμερίζομαι και προσυπογράφω κάποιες αψερωτήσεις της συναδέλφου Τρούιπερ. Ιδιαίτερα όταν αναφέρεται ότι αυτά τα 2,5 εκατομμύρια λέει είναι αναγκαία για να υπογραφεί η σύμβαση με ένα γραφείο αρχιτεκτόνων. Ταυτόχρονα όμως όταν οι πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας λένε ότι για την ρύθμιση, την πληρωμή για το κτίριο της, ε, του οίκου της ιστορίας θα χρειαστούν 21 λέει εκατομμύρια ευρώ και προφανώς τότε οι δαπάνες για τους αρχιτέκτονες τι θα είναι 10% του κόστους όλου του εγχειρήματο κτηριακά ίσως λοιπόν κάποια επεξήγηση επιπρόσθετα θα πρέπει να δοθεί από πλευράς του κυρίου Πέτερινγκ ή από πλευράς του εκπροσώπου του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάποιες επεξηγήσεις που πρέπει να δοθούν που είναι αναγκαίες για την αποσαφήνιση αυτού του θέματος. Για τις υπόλοιπες τεχνικές λεπτομέρειες η συνάδελφος Τρούπερ ήδη διατύπωσε πολύ σκόπιμες ερωτήσεις. Όμως εγώ εξακολουθώ να έχω μια αμφιβολία. Ένας από τους κύριους λόγους για τη λειτουργία για τον ε, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Προϋπολογισμό είναι το αίτημα της συγχρηματοδότησης εγώ ούτε και εγώ μπορώ να κατανοήσω πώς είναι δυνατόν τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή ακόμα και ο ίδιος ο Δήμος των Βρυξελών ή η ίδια η βελγική κυβέρνηση να μην ενστερνίζονται αυτό το εγχείρημα και να μην συνεισφέρουν με κάποια χρηματοδότηση για αυτό το εγχείρημα που έχει ενδιαφέρον και συμφέρον για όλους. Και επιπλέον στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρηματοδοτούνται εκδηλώσεις τεράστιας εμβέλειας ευρωπαϊκού χαρακτήρα δεν μπορώ να φανταστώ μια πιο σημαντική εκδήλωση ευρωπαϊκού χαρακτήρα από τη χρηματοδότηση ενό οίκου, ενό μουσείου ευρωπαϊκή ιστορία. Γι' αυτό θα έπρεπε να συμμετέχουν στον προπολογισμό αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χρηματοδότηση αυτού του εγχειρήματο. Ευχαριστώ. Mes Ευχαριστώ, Αγαπητοί συναδελφοί, είναι 11 η ώρα και πρέπει να ψηφίσουμε τώρα στις και έχουν ζητήσει έξω τώρα, έχουμε πάρα πολύ σημαντικές ψηφοφορίες, οπότε παρακαλώ μην μιλήσετε πάνω από ένα λεπτό και συμπαθάτε με γι' αυτό, αλλά Goran Farm. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε για αυτή την ε, παρουσίαση την ε, εξαιρετική και ευχαριστούμε και για όλη την ε, την τεκμηρίωση, τα έγγραφα που πήραμε, τόσο ώστε να δικαιολογείται αυτή η εκταμείευση. Τώρα μάθαμε περισσότερα από ό,τι πριν. Δεν είναι θέμα ε, τη δική μα επιτροπή αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή αυτή η υπόθεση και ιδίω μου άρεσε αυτό το οποίο αναφέρεται εδώ ότι θέλετε να επικεντρωθείτε στο θέμα τη ε, Ευρωπαϊκή Ιστορία μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ε, γιατί αλλιώ θα ήταν το θέμα πάρα πολύ πλατή, πάρα πολύ ευρύ Οπότε αυτό είναι και ο λόγο που το υποστηρίζουμε, ότι ακριβώ πρόκειται για το χρόνο, την περίοδο, τη φάση τη ολοκλήρωση. Αυτό είναι προσωπικέ απόψει και. Όμω, όμω, όμω, Πρέπει να σας πω ότι είναι επίσης πάρα πολύ καλή ιδέα να έχουμε μια αναφιερωμένη στρατηγική ε, για τους επισκέπτες. Αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παρά το ότι όπως και η κυρία Τρούπελ έχω και εγώ κάποιες ε, παρατηρήσεις όσον αφορά τα θέματα επιμελητίας, τα οργανωτικά και υπάρχουν κάποιες απαντήσεις που επιδέχονται ε, απαντήσεις είπαμε αυτή για την συγχρηματοδότηση και τη θεσμική προσέγγιση και εγώ έχω να σας πω το εξή Πρώτα-πρώτα ανεφέρθη εις το αρχικό ε, κείμενο των πυρογνωμών ότι πρόκειται εδώ πέρα για ένα, για ένα εξάρτητο φορέα. Μήπως μπορείτε να μας πείτε λίγο, λίγο παραπάνω τι εννοείτε όσον αφορά αυτό το, το, το, το χωριστό φορέα, το χωριστό ε, ίδρυμα. Όχι, δεν θα ανήκει στο οργανόγραμμά μας ούτως πεινά αλλά πέστε μας λίγο παραπάνω, διότι αυτό θα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να ξεκαθαριστεί αυτή η διαδικασία λήψη των αποφάσεων, διότι βέβαια είναι πάρα πολύ ε, ε, διφορούμε το θέμα μια που μιλάμε για περίοδο λιτότητας κάνουν όλοι ό,τι μπορούν αυτοί αύξηση του 1% όλοι θέλουν να κόψουν από τις διοικητικές δαπάνες ο κ. Φαραντής θα πει να μην γίνει καμία αύξηση ε, και επομένως τα πράγματα στριμώχνουν οπότε θα πρέπει να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων γιατί ένα πράγμα είναι η εκταμείευση, από την άλλη μεριά όμως πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει όσον αφορά την οριστική απόφαση. Θα γίνει ε, μια μεταφορά πόρων μέσα στον προπολογισμό των δικό μας ή χρειάζεται κάποιο άλλο είδους απόφαση για το σύνολο του οράματος αυτού. Επομένως, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πριν αυτές οι ερωτήσεις απαντηθούν, νομίζω ότι από πλευρά της, πολιτικής, ε, ομάδας μας θα ζητήσουμε μία ε, αναβολή. Όχι, όχι γιατί οι ερωτήσεις θα παρελθούν, αλλά πρέπει να μάθουμε τι θα γίνει, το κόστος του, του κτηρίου, όλα αυτά να ξεδεθούν πριν αποφασίσουμε. Ευχαριστώ. Γκόραν, ευχαριστώ. Πόρτας. σε ένα λεπτό σύντομα. Μου αρέσει αυτό το πρόγραμμα, το εγχείρημα για το μουσείο και επίσης μου αρέσει από ό,τι είδα το πρόγραμμα της εξωτερικής αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης αυτού του μουσείου. Είναι αναγκαίο αυτό το μουσείο πιστεύω και πιστεύω ότι τα κόστη που έχουμε εδώ μπροστά μας δεν είναι υπερβολικά και κυρίως έχουμε και άλλες μορφές εξοικονόμησης που μπορούν να αντισταθμίσουν αυτά τα κόστη στο μέλλον. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η κυρία Χέλγα Τρίπελ. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε από αλλού και έτσι λοιπόν θα πρέπει έτσι να το δούμε. Μία μόνη ερώτηση απομένει και κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με τον προλαλήσαντα θέλω να θέσω. Εγώ στη χώρα μου, στην Πορτογαλία, ένα γραφείο αρχιτεκτόνων, για παράδειγμα, το, το κόστος είναι 7 8% της συνολικής επένδυσης, αν το θυμάμαι καλά. 2,5 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν για μια τέτοια επένδυση, για 21 εκατομμύρια συνολικά που θα επενδυθούν, μου φαίνεται υπερβολικά υψηλή δαπάνη για τους αρχιτέκτονες. Αυτή είναι η μόνη ερώτηση που θα ήθελα να θέσω και να απαντηθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Μένουμε στην Πορτογαλία, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε αυτό το θέμα ήδη αποφασίστηκε, ήδη συζητήθηκε σε σχέση με τον προϋπολογισμό για το 2011. Τα κόστη επίσης βρίσκονται στην τεκμηρίωση για τα 52 εκατομμύρια ευρώ ή το κόστος τέλος πάντων του οίκου ευρωπαϊκής ιστορίας. Συγχαρητήρια για τις εξαιρετικές παρεμβάσεις που έγιναν εδώ, είτε από τον κύριο Πέτερινγκ, αλλά και από τον κύριο Αντιπρόεδρο Μαρτίνεθ Μαρτίνεθ. Και οι πληροφορίες για μας είναι σαφείς, απόλυτα σαφείς. Είναι αδύνατο προφανώς να επισέλθουμε στη συζήτηση λεπτομεριών τώρα όσον αφορά την καθαρή διαχείριση όλων αυτών. Και εμεί θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε όρου και θέση για κάτι επί του οποίου έχει ληφθεί απόφαση επί της ουσίας. Ένα δηλαδή πρωταρχικό σχέδιο. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ως σχέδιο αποφασιστεί, βρίσκεται υπό εξέλιξη, έχει δρομολογηθεί και μπορούμε να το συνεχίσουμε και στη συνέχεια να εξευρεθούν τα αναγκαία κονδύλια επενδύσεων για την εκτέλεση αυτών των έργων. Λαμβάνοντας υπόψη επίσης φυσικά και τους περιορισμούς που υπάρχουν από πλευράς προϋπολογισμού, από πλευράς κονδυλίων. Και αυτό είναι ένας όρος, μια προϋπόθεση που θα πρέπει να αναλυθεί όπως πρέπει στο μέλλον. Και έτσι δεν θέλω να προδικάσουμε κάτι, μια και έχει αποφασιστεί κάτι. Και έτσι έχουμε ήδη μια απόφαση του Κοινοβουλίου και έχουμε και τον προϋπολογισμό 2011 σχετικά. Ευχαριστώ. Merci, Κυρία Ολμάιερ, παρακαλώ. Πριν λεπτό το λόγο θα πρέπει να καλωσορίσουμε την κυρία Κρέσλη, η οποία τώρα μόλις μπήκε. Ίγκε. Ίγκε. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. C'était hier, c'était hier, mais comme elle l'a fêté depuis 24 heures, nous ne l'avons vu qu'aujourd'hui. Madame Monica Olmayer. Herr Vorsitzender, Sie hat... Et, κυρία Monica Ολμάιερ η ιδιαίτερη τιμή, Πρόεδρε, και για έναν Ευρωβουλευτή είναι κάτι ιδιαίτερο όταν έχει τα πεντηκοστά του γενέθλια και αυτά συνδέονται με τη νέα ρύθμιση της δημοσιονομικής, του δημοσιονομικού κανονισμού. Πραγματικά γιορτή και γενέθλια γιορταστικά αυτά. Πραγματικά εδώ αυτό είναι απόλυτα ε, σημαντικό. Τώρα για το, τον οίκο Ευρωπαϊκής Ιστορίας να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα για να αποσαφηνίσουμε τα θέματα των ποσών, των αριθμών, γιατί κάποια λανθασμένα ποσά υπήρχαν. 31 εκατομμύρια για την ανακαίνιση και την επέκταση. Το 2008 ξέρετε ότι πάντα εξετάζω τα ποσά ιδιαίτερα ξεχωριστά. Το 2008 στον, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών είχαμε την αγορά του κτηρίου Ίσμαν για 18,5 εκατομμύρια που είχαμε εγκρίνει. Τότε μόνο για την ανακαίνιση, αποκλειστικά ανακαίνιση, 18 εκατομμύρια είχαμε εγγράψει. Δηλαδή κατ' είναι η επέκταση που θα, θα χρειαστεί τώρα για τα 13 εκατομμύρια. Καταλήγουμε στα 31 εκατομμύρια λέει. Όμως τότε δεν είχε ποσοστοποιηθεί η επέκταση πόση θα ήταν, ποια θα ήταν. Έχουμε και ένα πρόσθετο έγγραφο το οποίο αναφέρει ότι για την εσωτερική, τον εσωτερικό εξοπλισμό μόνιμη έκθεση, ευέλικτες εκθέσεις, προσωρινές και εποχικές εκθέσεις και όλα τα συναφή απορρέουν από αυτά ότι 21 λέει εκατομμύρια συν χώροι συνεδριάσεων, χώροι για τη διοίκηση κτλ και συνολική παρουσίαση μεταξύ 2012-2014 3 εκατομμύρια επιμέρους δαπάνες. Ήθελα να παρακαλέσω αγαπητοί συνάδελφοι σήμερα να προβληματιστούμε και να δούμε ότι πρόκειται μόνο για μια μεταφορά κονδυλίων μόνο για τη μελέτη του αρχιτεκτονικού γραφείου για να μπορέσει δηλαδή να πληρωθεί αυτή η μελέτη και να συνεχίσει η διαδικασία του εγχειρήματος. Αν αρχίσουμε να θέτουμε ερωτήματα πού και θα έχουν τον τερματικό σταθμό τους λεωφορεία, πού θα παρκάρουν τα λεωφορεία και επιβαρύνουμε όλη αυτή τη συζήτηση διαδικαστικά. Αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε και σε τέσσερις εβδομάδες, στο μέλλον, υστερότερα. Να μην επιβαρύνουμε τέτοιου, με τέτοιου είδους διαδικαστικά ερωτήματα. Φυσικά κάπου, κάπου θα πρέπει να παρκάρουν, κάποιο θα είναι ο χώρο στάθμευσης, Θα ξέρουμε αυτά, ότι έχουμε και ένα γκαράζ άδειο κάτω στα υπόγεια το κτηρίου μας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι χώροι για τους και μπορούν να διατεθούν οι χώροι. Πολύ ωραία. Δεύτερο, πρέπει επίσης να προβληματιστούμε και για κάτι άλλο. Αν ένα τέτοιο εγχείρημα γίνεται τη σωστή χρονική στιγμή. Ισχυρίζομαι ότι τα προγράμματα ιστορίας και πολιτισμού ποτέ δεν γίνονται και δεν μπορούν να γίνουν στη σωστή χρονική συγκυρία. Διότι υπάρχουν πάντα άλλες ανάγκες, πιεστικές ανάγκες, κοινωνικές, οικονομικές και άλλες. Για μένα τίθεται το ερώτημα μόνο για τη μεταφορά ενός ποσού 2,5 εκατομμύρια εκατομμυρίων αυτό το θέμα να το παγώσουμε όπου μπορούμε στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα να εξετάσουμε να δούμε τι θα γίνει και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πληρώσει και εκείνη και να συνεισφέρει με τα έξοδα στο μέλλον τώρα όμως αυτά τα 2,5 εκατομμύρια ως μεταφορά να επιβαρυνθούν με άλλες επιβαρύνσεις ως όρους και προϋποθέσεις πιστεύω ότι το πρόγραμμα αυτό ποτέ δεν θα είναι υλοποιήσιμο και εφικτό κυρία Τρούπερ του Αγίου ποτέ θα το αναβάλουμε στις ελληνικές καλένδες. Να μην το επιβαρύνουμε λοιπόν, γιατί στο Συμβούλιο 27 κράτη-μέλη θα πάρουν τον λόγο και θα πρέπει να ομοφωνήσουν και τι θα γίνει μετά. Λοιπόν, γι' αυτό να γίνει η προσπάθεια να συνεισφέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι άλλοι, να το δούμε αυτό. Αλλά να μην εξαρτηθεί η μεταφορά αυτού του κονδυλίου 2,5 εκατομμυρίων από αυτού του όρου και προποθέσει. Και για τα 31 εκατομμύρια το κόστο του αρχιτεκτονικού γραφείου βρίσκεται μέσα στα όρια όρια των μελετών που, ε, που πληρώνονται στις χώρες μας ε, με ανάλογο τρόπο. Αυτό εφόσον απαντηθεί έτσι μπορεί να προχωρήσει. Δεν υπάρχει κάποιο αρνητικό στοιχείο λοιπόν να επιβαρύνει αυτή τη μεταφορά. Συγγνώμη Πρόεδρε, ολοκληρώνω, δεν θα χρονοτριβήσω. Παρακαλώ αυτή τη μεταφορά κονδυλίου, αυτή τη μεταφορά πόρων να την εγκρίνουμε. Και όλα τα θέματα που εκκρεμούν κατά το επόμενο εξάμεινο να τα εξετάσουμε για να μην τώρα εδώ επιβαρύνουμε τα πράγματα. Vladimir. Ευχαριστώ, Βλαντίμη. Πολύ σύντομα, παρακαλώ. Ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, από πλευρά μου, σε σχέση με την εισήγηση για τον προπολογισμό, ήδη τότε πρέπει να πω ότι είχαμε συμφωνήσει ότι αυτή η μελέτη ήταν εντάξει και όλοι μας είχαμε συμφωνήσει ότι αυτή η επένδυση θα έπρεπε να γίνει μόνο που ένα ξεχωριστό κονδύλιο δεν το δημιουργήσαμε τότε επειδή θέλαμε προηγούμενα να υπάρξουν όλα τα επακριβή ποσά. Και για πρώτη φορά, μια και αναφέρθηκαν κάποια τέτοια στοιχεία, πρέπει να καθορίσουμε για το μέλλον το εξής. Ας μην κάνουμε περαιτέρω μεταφορές. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα πρόγραμμα δράσης πότε θα είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες για να μπορέσουμε έτσι να δράσουμε διότι κάποια μέρα αυτό το τρίγωνο θα πρέπει να λειτουργήσει. Αυτά τα τρία κέντρα δηλαδή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κέντρο Πληροφόρησης και ο Οίκος Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Σε αυτό το τρίγωνο συσχετισμού πρέπει να αποφασίσουμε αν αυτός ο Οίκος Ευρωπαϊκής Ιστορίας θα χρησιμοποιείται και το Σαββατοκύριακο για να υπάρχει πιο αποτελεσματική χρήση του. Θα είναι μια μόνιμη έκθεση αυτή ή θα πρόκειται για μια περιφερόμενη έκθεση ή εποχική έκθεση ή για τις μελλοντικέ δραστηριότητες πώς θα διαμορφωθούν και πώς θα αλλάζουν διότι αν αυτά αλλάζουν ετήσια θα έχει υπερβολικό κόστος μια τέτοια αλλαγή. Πρέπει όλα τα στοιχεία να τεθούν επί τραπέζης για να μπορέσουν να εκτιμηθούν. Δεν είναι δυνατόν να εγκρίνουμε μια μεταφορά κονδυλίων και μετά να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Συμφωνώ ότι με αυτό που είπε η κυρία ε, Τρίπερ, ότι η πόλη των Βρυξελών, ο Δήμος των Βρυξελών πρέπει να αποτελέσει εταίρο μας. Και αυτό θα ήταν υποφελές για τις Βρυξέλλες. Πολλοί επισκέπτες έρχονται στις Βρυξέλλες, τουρίστες και κανένας φυσικά δεν είναι δυνατόν να μειώσει αυτό το προτέρημα για μας ότι εμείς είμαστε οι πρώτοι που αποφασίσαμε κάτι τέτοιο. Ο Ανδρέας παρακαλώ. Thank you, Yeah, η κυρία, Ανδρέας, ε, κυρία Ανδρέας, ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσαφιλιστεί ποιος είναι ο κύριο, ποιος έχει την κυριότητα αυτού του κτηρίου. Διότι αν υπάρχουν ε, κόστη όσον αφορά τη μίσθωση, έστω και σε σχέση με την Επιτροπή, θα ήθελα να δοθεί απάντηση ποιος θα έχει την κυριότητα αυτού του κτηρίου. Εσείς κύριε Πέτερν είπατε ότι θα είχαμε πριν ξεκινήσει η λειτουργία αυτού του ε, κτηρίου ευρωπαϊκής ιστορίας 16 λέει εκατομμύρια ευρώ θα ήταν ε, το πρώτο κόστος. Δεν έχουμε όμως πληροφορίες για τις τρέχουσες δαπάνες. Ακόμα και όταν λέει η κυρία Ολμάιερ να εγκριθεί η μεταφορά κονδυλίων για την αρχιτεκτονική μελέτη, διαφωνώ απόλυτα να λάβουμε μια απόφαση με αυτόν τον τρόπο προτρέχοντας χωρίς να έχουμε υστερότερα στοιχεία στη διάθεσή μας. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για τέτοιου είδους δαπάνες, ακόμα και αν χρηματοδοτείται με άλλες δράσεις. Την ιστορία μπορεί να, την, ε, να προσφύγει κανείς στη βιβλιογραφία ή ε, σε ε, αντίστοιχες μελέτες. Γιατί χρειάζεται λοιπόν ένα ξεχωριστό οίκο ευρωπαϊκής ιστορίας η Ευρώπη. Ακόμα και σε μια περίοδο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο συγκυρίας, προσβάλλουμε τους πολίτες της Ευρώπης όταν κάνουμε πρόσθετες δαπάνες σε μια περίοδο περικοπών στους εθνικούς προϋπολογισμούς, σε μια περίοδο αυστηρής λιτότητας να κάνουμε τέτοιες δαπάνες. Επίσης αμήχανο είναι δημιουργία μηχανία να μπορεί το Κοινοβούλιο να προχωρεί μόνο του στην εκτέλεση ενό τέτοιου έργου χωρί συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή του Συμβουλίου. Αυτή θα έπρεπε να ήταν η αφετηρία, να συμμετάσχουν όλα τα θεσμικά όργανα κατά αναλογία μεταξύ τους. Εμείς δεν θα εγκρίνουμε αυτή τη μεταφορά. Ούτε οποιοδήποτε άλλο κόστος το οποίο θα συνεπάγεται η δημιουργία αυτού του οίκου ευρωπαϊκής ιστορίας. Ευχαριστώ. Ο αγορητή είναι η Γιούτα. Χάουκ. Η κυρία Χάουκ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, προσέξτε, ευθύ εξ αρχή το Συμβούλιο και την Επιτροπή να τους είχαμε στο πλευρό μας ως εταίρους. Δεν το εκτιμώ αυτό. Ξέρουμε τι γίνεται όταν προσπαθούμε με το Συμβούλιο να ομοφωνήσουμε ή να καταλήξουμε σε κάποιους συμβιβασμούς. Ας αφήσουμε τα χέρια μακριά από το Συμβούλιο. Είναι προειδοποίησή μου. Αλλά όσον αφορά αυτά τα, αυτούς τους δισταγμούς, αυτές τις επιφυλάξεις, αυτό συσχετίζεται με το ότι εδώ στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και εγώ δεν αντιμετωπίζω το ίδιο το εγχείρημα δεν έχουμε την εντύπωση ότι ξέρουμε με τι πράγμα ασχολούμαστε και ποιε θα είναι οι τελικέ επιπτώσει. Ετήσιο κόστο όσον αφορά τι δαπάνε, για παράδειγμα. Εδώ στην 6, σελίδα υπαριθμών 6, για πρώτη φορά έχουμε τρέχουσε δαπάνε. Running costs όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό. 7, 2-9 εκατομμύρια ευρώ αναφέρονται. Εντάξει, αλλά για το προσωπικό δεν ξέρουμε τίποτα. Δαπάνε για τα στελέχη. Ναι, μεν αναφέρονται κάποιε θέσει που θα χρειάζονται, αλλά κανεί δεν μα λέει ποιοι θα είναι οι μισθοί και ποιο θα είναι το συνολικό μισθολογικό κόστο. Υπάρχουν προβλήματα λοιπόν εδώ. Αν θέλουμε να έχουμε μια σαφή εικόνα για όλα αυτά. Θα ήταν θετικό για μας που είμαστε αρμόδιοι για θέματα προϋπολογισμού δημοσιονομικά. Για μας θα ήταν απλούστερο το θέμα. Δεν αντιμετωπίζω το θέμα του εγχειρήματο ως θέμα αρχή, αλλά θα διευκόλυνε αν είχαμε αυτά τα στοιχεία για να εγκρίναμε. Ευχαριστώ. Ό,τι βλέπετε, η συζήτηση είναι πάρα πολύ πλούσια, πάρα πολύ ζωντανή, ένα σωρό όμως εγώ είμαι υποχρεωμένος εδώ να βάλω τελεία, διότι έχουμε τις ψηφοφορίες που δεν μπορούμε να τις αναβάλουμε γιατί πρέπει, πρέπει η Επιτροπή μας να είναι έτοιμη για να ληφθούν οι αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν την επόμενη εβδομάδα ή στην Ολομέλεια. Όμως υπενθυμίζω κάτι που είπανε πολλοί συνάδελφοι ότι το Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια και συγκεκριμένα η Επιτροπή των Προπολογισμών εστήριξαν ε, από είπαν αρχή την υπόθεση αυτή το είπε η συγκεκριμένη επιτροπη των Ανδρέας όλοι, όλοι, όλες τις πολιτικές ομάδες Οπότε αυτό ο οίκο της ευρωπαϊκής ιστορία που είναι κάτι που το ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε πρώτη φάση το χρηματοδότησε ακριβώς όπως είπε ο κύριος Μαρτίνες Μαρτίνες, ο πρόεδρος ε, το ε, το έκρινε και τώρα ω Επιτροπή των Προπολογισμών πρέπει διαδοχικά να λάβουμε δύο αποφάσει. η πιο επίγουσα αφορά το πώ θα αποδείμουν αυτό, το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων σε σχέση με αυτή την πίστοση που είχε εγγραφεί στον προσμό της χρήσης 2011 και έχει μπει στο αποθεματικό ε, με την επιφύλαξη του ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιε διευκρινήσει για το κτίριο κλπ. Και όσον αφορά την διαδικασία. Τι Συνέχεια δε έχουμε ε, το κείμενο Φερνάντες οπότε θα πρέπει να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις με το Προεδρείο ποιο ακριβώ είναι το ποσό του πιθανή γραφεί ή στον προηγούμενο του 2012, 12 δεν είναι πρόεδρο, όχι 11, 12 για τη χρήση 12 όσον αφορά κάποιε τέτοιε διευκρινήσει. Αυτά στον προπολογισμό. Τώρα, θέτω ει τον εισηγητή το εξή. αν κατάλαβα καλά τι έχει να μα πει, ή εισηγήτρια τέλο πάντων, ε, διαπιστώνω ότι υπάρχουν κάποιες πολιτικές ομάδες όπως οι σοσιαλιστές οι οποίοι θέλουν να υπάρχουν κάποιες διευκρινήσεις πριν γίνει η εισηγητρια τελο παντων διαπιστωνω οτι υπαρχουν καποιε πολιτικε ομαδε οπω οι σοσιαλιστε οι οποιοι θελουν να υπαρχουν καποιε διευκρινησει πριν γινει η ψηφιση όσον αφορά την εκταμείευση των χρημάτων. Εάν επομένω θεωρείται, ε, θεωρεί η συγκίτρια ότι χρειάζεται κάποιε τέτοιε πριν πάμε για την ψηφοφορία για την πληρωμή του ποσού, σα προτείνω να αναβληθεί η ψηφοφορία. Και επίση ε, βλέπω ότι κανεί δεν αντιτίθεται. Όμω ορισμένοι χρειάζονται. Πριν δώσετε το πράσινο φω, αυτέ τι διευκρινήσει. Και προτείνω την αναβολή. 15 Μαρτίου. Και μέχρι τότε. Πρώτον, οι να είναι συντονισμένοι με μια ομάδα συναδέλφων κ. Φερνάντε και κ. Αλμάγερ οι οποίοι έχουν ε, αναλάβει την υπόθεση των ε, κτηρίων μαζί με την Έλγα να έρθουν σε επαφή με τους άλλους συναδέλφους και να ε, ξεκαθαριστεί ποια ερωτήματα θέλουν να απάντησε ούτως ώστε να γίνει εκταμείωση των πόρων. Διότι ακριβώ φίλοι ετέθεσαν πάρα πολλά ερωτήματα ε, όσον αφορά τη, τη μακρόπνα ε, προοδευτική, το, το κόστο λειτουργία του κτηρίου κλπ. κλπ. Όμω δεν είναι αυτό το οποίο τώρα πρέπει να, να απαντηθεί. Κάποια άλλα θα πρέπει να ούτω ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε το πράσινο φω για την πληρωμή. Οπότε σα προτείνω αυτή η μικρή ομάδα των τριών εκπροσώπων της ε, Επιτροπής των Προπολογισμών να έρθει μετά τη συνάντηση αμέσως σε επαφή με αυτούς που έχουν αναλάβει την υπόθεση του, του οίκου της ε, ιστορίας Ευρώπης και έτσι να έχουμε ρωτήσει απαντήσεις και εγγράφους και στην επόμενη συνάντησή μας 15 Μαρτίου τότε να είμαστε έτοιμοι για την ψηφοφορία όσον αφορά την πληρωμή. Οπότε, πια, μπορεί να ξεκαθαριστεί η θέση μας όσον αφορά τον προπολογισμό 2012. Μια τεχνική επισήμανση μόνο. Θα ακολουθήσει μια ξεχωριστή πληροφόρηση με όλε συνολικά τι λεπτομέρειε όσον αφορά τα κτίρια και όλα τα συναφή. Θα έρθουν όλα αυτά υστερότερα, εκτό από τη μετα... από τη μεταφορά. Με τη μεταφορά κονδυλίων δεν θα ξεκινήσει να δρομολογείται η πλήρη εκτέλεση αυτού του εγχειρήματο. Ευχαριστώ. Oui, συμφωνούμε. Χέλγα, σας ε, ικανοποιεί αυτή η λύση. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Τη βρίσκω σωστή αυτή τη λύση, γιατί τώρα δεν έχουμε πια άλλο χρόνο. Παραμένουν πολλά ερωτήματα που εκκρεμούν και γι' αυτό συμφωνώ με την πρότασή σας. Να αναβληθεί η ψηφοφορία. Μέχρι τότε θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε όλα αυτά τα θέματα μέχρι τέλη Μαρτίου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, βλέπετε ποια είναι η δική μας προδιάθεση, Πρόεδρε. Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση. Πρέπει να διακόψω τη συζήτηση. Αν τη διακόψω και ψηφίσουμε, εσείς δεν θα είναι δυνατόν να απαντήσετε και να θέλετε ως άνθρωπος όλες τις ερωτήσεις που τίθεται. Ωστόσο διαπιστώνεται το σημαντικότερο. Υπάρχει πολιτική στήριξη από πλευρά Επιτροπή Προπολογισμών και θεωρούμε όλοι ότι υπάρχει υποχρέωση να ε, έχουμε αποτέλεσμα. Θα σα βοηθήσουμε ω Επιτροπή Προπολογισμών. Υπάρχουν κάποια διευκρινιστικά που πρέπει να τα αποσαφηνίσουμε. Θα γίνουν αυτά ε, μέσα στο επόμενο 15 και μετά θα προχωρήσουμε στην πληρωμή. Και με τον κύριο Φερνάντε και το Προεδρείο θα δούμε τι ακριβώ θα γίνει για το 2012. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Θα συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι μπορούμε να ψηφίσουμε, να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Έχουμε τις ψηφοφορίες και σας προτείνω να ξεκινήσουμε με το σημείο 15 της σημερινής διάταξης. Έκθεση του συναδέλφου κ. Φερνάντες. Το συζητήσαμε την περασμένη φορά. Έχετε λάβει όλοι τον κατάλογο των ψηφοφοριών. Απλώς κοιτάξτε μήπως υπάρχουν περισσότεροι από το ΕΛΚ ή από τους Πρασίνους μεταξύ άλλων. Διότι σε αυτή την επιτροπή μόνο το ΕΛΚ εργάζεται, έτσι. Και όλα αυτά για να ξέρω αν έχω το δικαίωμα να ψηφίσω εγώ ή όχι. Τέλος πάντων. Όλοι έτοιμοι. Τέλεια. Τροπολογία 1. Αιτιολογική σκέψη G. Κύριος Άλβαρο. Ο εισηγητή είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγκρίνεται ομόφωνα. 2. Βόγκαν. Ο εισηγητή υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν υπάρχουν αποχέ. Εγκρίνεται. Τρία, κύριο Άλβαρο. Κατά ο εισηγητή. Υπέρ. Πρέπει να μετρήσουμε. Κατά. Μπορώ να ψηφίσω. 15 ε, και 16 είστε κατά, κυρία μου. Πολύ ωραία. Ε, Αλλάζετε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. madame, je, salue votre courage politique. Ε, χαιρετίζω την πολιτική σας τόλμη. Τέσσερα. Έλε, Κατά γιατί... Πέρ. Και πάλι πρέπει να μετρήσουμε. Έχουμε και τα μηχανήματα, έχετε το τις κάρτες σας. Για να μετρήσουμε για αυτή την ψηφοφορία και την επόμενη φορά θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Bon, alors, euh, levez les bras Παρακαλώ, σηκώστε ολόκληρο το χέρι, όσοι είστε υπέρ. Δεκαεπτά, τέλεια. Υπέρ, κατά. Ψήφι κατά. 6, 7, vote 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Χαχά. Απορρίπτεται η τροπολογία. 5. Βόγκαν. Υπέρ ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6. Βόγκαν. Υπέρ ο συγκεκριτής. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7. Άλβαρο. Υπέρ, ο συγκεκριτής. Υπέρ. Πολύ. Κατά. Κανείς. Αποχές. Μία. 8 προφορική τροπολογία του κυρίου Άλβαρου. Συνάδελφε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λυπούμε που μέσω προφορικών τροποποιήσεων πρέπει να προχωρήσουμε. Αλλά μια και ο πίνακα ψηφοφορία voting list ήρθε σε εμά όταν βρισκόμαστε στην Κοπενχάγη ω κοινοβουλευτική ομάδα και δεν είχαμε συνάντηση σκιωδών εισηγητών, λυπούμε για την προφορική τροποποίηση. Αναφέρεται στην παράγραφο 3 ε, ελαφρά αλλαγή. Οι αρχές της χρηστής διακυβέρνηση και διαχείριση για τα οικονομικά αναφέρονται η λογοδοσία, accountability, δεν αναφέρεται εδώ ρητά. Υπό το πρίσμα λοιπόν και το πνεύμα της accountability, λογοδοσίας που θέλουμε να ενταχθεί εδώ. Αυτό αποσαφήνιση μια και δεν βρίσκεται στο άρθρο 27 η λογοδοσία, accountability, γι' αυτό θέλουμε να είμαστε υπό το πνεύμα της λογοδοσίας, in the spirit of accountability, θέλουμε να υπάρξει τροποποίηση, προσθήκη δηλαδή. Ελπίζω δεν θα υπάρξουν ενστάσεις για να μην γίνει δεκτό αυτό. Ευχαριστώ. Je comprends Βλέποντας το χαμόγελο του εισηγητού, καταλαβαίνω ότι είναι υπέρ αυτής της προφορικής τροπολογίας. Πολύ ωραία. Ψηφίζουμε για την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ομοφωνία. Για το πνεύμα του κυρίου Άλβαρο. Εννέα. Βόγκαν Φέρμ. Δεν αρέσει πολύ στον εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Προφανώς πλειοψηφία. Αποχές σε μειοψηφία αριστερά. Δέκα. Και πάλι κατά ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Πολύ. Αποχές μία περίπου ίδια πλειοψηφία. Απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση. 11. Άλβαρο. Δεν αρέσει τον εισηγητή. Υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Le vote électronique est ouvert. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχω δικαίωμα να ψηφίσω έτσι, δεν είναι πολύ συνάδελφοι από το ΕΛΚ. Ωραία. Δεν έχετε κάρτα και είστε κατά. Α, όχι, είστε υπέρ. Πέρας. 18 υπέρ. Ο κύριος Αίντερ 19. Εγκρίνεται. 13 όχι, με συγχωρείτε, αυτό ήταν το 11. Όχι, ήταν το 12. Ε, 12 ε, τώρα. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Πλειοψηφία κατά. Απορρίπτεται. 13 έλες. Υπέρ ο εισηγητής. Υπέρ. Όλα τα χέρια σηκώθηκαν. Κατά. Κανείς. Αποχές. Κανεί. Μπράβο, Τζέιμ. Ομοφωνία. 14. Ο εισηγητή είναι υπέρ. Υπέρ. Πολύ κατά. Ο κύριο Άλβαρο. Και μερικοί ακόμα. Δημοκρατία. Έχουμε αποχέ. Εγκρίνατε. 15. είδατε. 16. Αντάμ. Αμπάντρικε. Υπέρ ο εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ αποχές. Εγκρίνεται. Παρά την ψήφο της Έλγα. 17. Υπέρ ο συγητής. Υπέρ. Και η ΕΛΓΑ είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται ομόφωνα. Και πάλι και τροπολογία στο 18. Να προσθεθούν redeployment and training. Υπέρευσε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται ομόφωνα. Έχουμε τώρα συμβιβαστική α, κεφαλαίο α, του εισαγητού. Ο κύριος Βόγκαν θέλει το λόγο από αυτού. Όχι, ναι. Συνάδελφοι, αρχικός, η τροπολογία α μου είχε παρουσιαστεί από τον εισηγητή σε μια άλλη μορφή. Τώρα, μετά από συζητήσει, ε, συμφωνήσαμε σε μια νέα μορφή. Τη είναι αρκετά μακροσκελή, θα τη διαβάσω. Ο εισηγητή νομίζω ότι είναι υπέρ. Ελπίζω ότι θα το δεχτούν οι συνάδελφοι ω νέα τροπολογία Α. Συμβαστική Α. Σα ευχαριστώ. Κύριε Άλβαρο, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγγλικά θα τα πω. Σας ευχαριστώ πολύ για το νέο σχέδιο, νέα διατύπωση για την συμβαστική τροπολογία. Αυτό δείχνει ιδιαίτερα ότι θα έπρεπε ουσιαστικά να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Εκείνο όμω το οποίο δεν κατανοώ ακόμα είναι γιατί ουσιαστικά οι δύο μεγαλύτερε ομάδε ε, που ήταν υπέρ τη αύξηση ε, τη ε, επιδότηση γραμματεία τώρα είναι κατά των πρόσθετων κονδυλίων για γραφεία. Όταν έχουμε περισσότερου βοηθού χρειαζόμαστε περισσότερου χώρου γραφείων. Μερικά πράγματα δεν τα κατανοώ. Πώ είναι δυνατόν να γίνεται κάτι τέτοιο λοιπόν. Αυτό είναι απώλεια συνεκτικότητα και συνάφεια. Ουσιαστικά αφορά την προηγούμενη, το, ε, το προηγούμενο συμβιβασμό στην τροπολογία. Ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε εσεί οι Εντάξει, αυτό είναι όμω εξήγηση ψήφου. Και είναι εξήγηση θετική ψήφου. Λοιπόν, ψηφίζουμε για την ε, τροπολογία Α, τη συμβιβαστική Α, υπέρ. Κατά. αποχέ Εγκρίνεται. 19. Καταπίπτει. 20. Εσύ υπέρ υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία. Η Χέλγα. Και πάλι. Εγκρίνεται. Συμβαστική Β και Σ. Τις ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται και η B και η C. 21, 23, 25, 28 εκπίπτουν. 22. Χέλγα Τρίπελ. Ο εισηγητή είναι υπέρ. Υπέρ. Μεγάλο ενθουσιασμό, Κατά. Κανεί, Αποχέ. Ομοφωνία. Μπράβο Χέλγα. 24. Άλβαρο. Εισηγητή υπέρ. Υπέρ. Κατά. Η κυρία Ανδρέασεν. Τρεις κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D του εισηγητού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26 και 27 καλύπτονται. 29 μάνκα. Υπέρ ο εισηγητής, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται ομόφωνα. Μπράβο, Βλάντιμιρ. 30. Βόγκαν Φέρμ. Αποσύρεται. 31. Βλάντιμιρ. Ο εισηγητή είναι υπέρ, υπέρ. Κατά. Μία ψήφο κατά. Τρει ψήφοι κατά. Αποχέ. Δύο. Εγκρίνεται. 32. Βλάντιμιρ. Ο εισηγητή είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Τέσσερις ψήφοι κατά. Αποχές, όχι. Εγκρίνεται. 33 έλες. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Κατά εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Πλειοψηφία. ξεφανίστηκε το πρώτο τμήμα. Πρόεδρε, μπορώ να κάνω μια προφορική τροπολογία για το δεύτερο τμήμα, αφού Χάσαμε το πρώτο. Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει μια τέτοια έκθεση ω 30, 30 Ιουνίου του 2011. Ο εισηγητή τι γνώμη έχει για την προφορική τροπολογία που θα συμπληρώσει το δεύτερο τμήμα. Υπέρ ο εισηγητή. Υπέρ. Για την τροπολογία όπω τροποποιήθηκε με την προφορική τροπολογία του Τζέιμ. Κατά. Μία ψήφο κατά. Αποχέ. Μία. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. Όπω το συμπλήρωσε ο προφορικό ο Τζέιμ. 34. Αποσύρεται και η πόρτα. 35. Όχι. Όμω ο εισηγητή δεν το θέλει. Δεν τη θέλει η τροπολογία. Υπέρ. Ο κύριο Πόρτα και η κυρία Ανδρέασεν. Περίεργη συμφωνία. Αξιοσημείωτη. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38. Άλβαρο. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ. Μερικοί. Κατά. Πολύ. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 Βλάντιμιρ Μάνκα. Ε, υπέρ ο συγκεκριτής υπέρ. Κατά. Είναι φιλελεύθερη. Όμω είναι μειοψηφία, οπότε ο Βλάντιμιρ κέρδισε. Αποχέ, ωραία. 40, Άλβαρο. Αυτή τη φορά ο συγκεκριτή είναι υπέρ, υπέρ. Διευκολύνουμε έτσι τα πράγματα. Κατά. Κανείς. Αποχές. Εγκρίνεται ομόφωνα. Μπράβο στον Αντιπρόεδρο Άλβαρο. 41. Προφορική τροπολογία για την έγκριση του τίτλου. Υπηρεσία αξιολόγηση ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Υπέρ, τι υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται ομόφωνα. 42. Δεουρκίθα. Ισπανικό είναι. Κυρία, με συγχωρείτε. Εσείς είστε κυρία μου. Με συγχωρείτε. Της κυρίας Δεουρκίθα, λοιπόν. 42. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές πλειοψηφία κατά. Με λυπούμε κυρία Μό. 43. Εδώ η συγκεκριτής είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44. Κατά ο συγκεκριτής. Υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. 45 κατά ο Απορρίφθηκε η προηγούμενη, δεν ακρίθηκε. 45 κατά ο υπέρ. Μόνο οι σοσιαλιστές. Κατά. Όλοι οι υπόλοιποι. Αποχές απορρίπτεται. 46 τα ίδια, ο εισηγητής κατά. Υπέρ. Κατά Απορρίπτεται. 47 τελευταία τροπολογία της κυρίας Δεορκίθα, κατά της και πάλι, υπέρ. Λίγη παραπάνω. Τι ωραία, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, κυρία Δεορκίθα. Ε, ε, ε, ναι, ναι, έχει την κάρτα της, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε, ψηφίστε, δεν ψήφισαν όλοι. Κρίμα, δεν προλάβατε. Πέρασε τη ψηφοφορία. 16 υπέρ, 19 κατά. Απορρίπτεται. Ορίστε. Θέλει να πει κάτι ο για την τελική ψηφοφορία. Όχι, μια τροπολογία τεχνικού χαρακτήρα. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Για το 23. δεν είναι 86 εκατομμύρια 186 εκατομμύρια ευρώ μάλλον αλλά 149,6 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι είναι τεχνική τροπολογία. Ε, ναι, είναι ένα μικρό σφαλματάκι, μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Είναι λίγο τεχνικό το θέμα. Δεν φαίνεται να υπάρχουν διαφωνίες για αυτή την τεχνική τροπολογία. Τελική ψηφοφορία. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 34 υπέρ, 1 κατά, μία εποχή. Συγχαρητήρια. Στον εισηγητή. Ωραία, λοιπόν, αυτό το φέραμε σε αίσιο πέρας. Τώρα, πρέπει να ψηφίσουμε point 16. Sur le point 16. Για το 16 τώρα. 16 και 17. Ε, προβλέπεται να ψηφίσουμε. Όμως να δώσω το λόγο εις, την εισηγητρία, την Σιδονία, η οποία θα μας εξηγήσει γιατί προτείνει να μην ψηφίσουμε. Ε, κολεζάνκι, ε, ε, Sprawa dotyczy Funduszu Solidarności, o którym πρόκειται για αυτό το Ταμείο Ελεγγύης. E, Τα συζητήσαμε. Και λέγαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτό, αυτή η υποστήριξη, η χρηματοδότηση από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό αφορούσε τις χώρες που επλήγησαν πέρυσι από τις πλημμύρες. Η δε έκθεσή μου δεν θα έπρεπε σήμερα να ψηφιστεί και να σας εξηγήσω. Να σας εξηγήσω. Μας ενημέρωσαν ότι ορισμένα κράτη-μέλη δεν επιθυμούν να υποστηρίξουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε ε, υπάρχει επομένως μία αντίσταση από τα κράτη-μέλη. Και με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνουμε, διαπιστώνω ότι η Ουγγαρία ως Προεδρία προσπαθεί κάτι να κάνει στο Συμβούλιο, να κινηθούν τα πράγματα, όμως ε, έχουμε εδώ πέρα εμπλοκή στο Συμβούλιο, γιατί επί της αρχής φυσικά και πρέπει να εκταμεθεί το ποσό από το Ταμείο Ελληνικής, όμως για τεχνικούς λόγους δεν μπορούν να ανεβρεθούν τα κονδύλια. Επομένως, περιμένουμε να μάθουμε τι θα γίνει στην Κορεπέρ. Δεν ξέρουμε τίποτα ακόμα. Την επόμενη εβδομάδα κάτι θα προκύψει. Οπότε πασχίζουμε να βρούμε μια άλλη λύση. Ακόμα δεν ξέρουμε πάντως τίποτα. Επομένως, δεν υπάρχει κάτι που το οποίο να ψηφίσουμε τώρα. Δεν ξέρω, Πρόεδρε, τι, τι πρεσβεύεις. Μήπως πρέπει να μιλήσουν με το Συμβούλιο και να μας πούνε σε ποια φάση βρίσκονται ή να μας πει ξέρω εγώ η Κομισιόν τι αν είχε αλλάξει τίποτα από τα αρχικά σχέδια και έτσι να προχωρήσουμε προς μια λύση. Και επομένως τα λεφτά αυτά να πληρωθούν από το Ταμείο Ελληνική. Ευχαριστούμε κυρία Συγγετρία. Εγώ επ' αυτού σας πληρώνω λέει ο Πρόεδρος. Πάρα πολύ ξεκάθαρα μας εξηγήσατε πώς έχουν τα πράγματα από πολιτική και όπως έγραψε το πρωί κάποιο δημοσιογράφος ε, δεν πρόκειται για, για, για ε, την πρώτη αψημαχία. Θα ακολουθήσουν και άλλες όσον αφορά τους επόμενους μήνες ε, μεταξύ των, των διαφόρων συναρμοδίων ε, θεσμικών οργάνων. Από τη μία το Συμβούλιο και από την άλλη η υπόλοιπη όσον αφορά τις πιστώσεις των πληρωμών που εκρίθησαν πέρυσι και προβλέπεται αυτό το σημείο να ενταχθεί στην μεσή διάταξη του τριγωνικού διαλόγου της 31ης Μαρτίου οπότε εγώ σας προτείνω αυτή η συζήτηση να γίνει εκεί, στον τριγωνικό διάλογο, στον τριμερή διάλογο. Και αναλόγως τι θα προκύψει να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε οπότε. Θα φτάσω στον το 18 και το θέμα 18 κλείνει εδώ. Και επομένως αυτό ολοκληρώνει και την ε, δουλειά μας επί της εκθέσεως Μπέγγε και συνεχίζουμε τις ε, ψηφοφορίες. Πρωτόκολλο για ελληνική συμφωνία με τις Κομόρες. Αυτό αφορά τον κύριο Αλφόνης, ο οποίος δεν είναι εδώ. Ε, μία και μόνη ψηφοφορία θα γίνει. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ, ζητεί ο εισηγητής. Είναι, ποιος είναι υπέρ αυτής της αλληλευτικής συμφωνίας με τις Κομόρες. Ευχαριστώ. Ποιοι είναι κατά. Αντρέας. Αποχές δεν έχουμε. Και επομένω η Ελευθερική Συμφωνία με τι Κομόρε εγκρίνεται. Και συγχαρητήρια προ τον κύριο Αλφόνση, αν και λείπει. Και τώρα ή στην συνέχεια θα δούμε τι γίνεται με κάποιες εκτανιεύσεις, μεταφορές ε, κονδυλίων. Η Σιδόνια τώρα είχε ένα θέμα σχετικά με ένα άλλο σημείο και θα μας πει τώρα τι γίνεται όσον αφορά τις αιτήσει μεταφοράς των πιστώσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή η μεταφορά πόρων είναι πολύ σημαντική, διότι πρόκειται για ένα μεγάλο ποσό. Και στην τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής συζητήσαμε το γεγονός ότι συσχετίζεται με αυτό το συνολικό ποσό σε σχέση με, την, με μια ιδιωτική εταιρεία και αποφασίστηκε ότι θα έπρεπε να πληρώσει η εταιρεία αυτό το κονδύλιο εξέτασα αυτό το θέμα σε βάθος και το συζήτησα και σε λεπτομέρειες. Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει κατά της νομολογίας, κατά της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Για να συντομεύσω, πρόκειται για μια πολυετή αντιπαράθεση για την κυριότητα ενός προγράμματος λογισμικού ε, software για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και για κάποιες αλλαγές σε σχέση με αυτό. Αυτή τη στιγμή αμφισβητεί την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγοντας ότι ερμηνεύει με διαφορετικό τρόπο την κατάσταση των πραγμάτων όπως έχει διαμορφωθεί και γι' αυτό ασκούν προσφυγή κατά της απόφασης. Όμως πρέπει να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως ε, αρχικά προβλεπόταν σε σχέση με την αντιπαράθεση που είχε παρουσιαστεί στο Συμβούλιο. Έχασαν και έτσι πρέπει να πληρώσουν και σε σχέση με πρόσθετες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά. Παρόλα αυτά όμως υπό το δικό μου πρίσμα προσωπικά μπορώ να πω ότι σε σχέση με το σύστημα όπως έχει διαμορφωθεί από αυτήν την εταιρεία και την αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα πράγματα δεν είναι τόσο προφανή διότι ποτέ δεν είχαν υποβληθεί γραπτός οι αμφιβολίες που υπήρχαν σε σχέση με θέματα ή θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όταν υπήρχε, υπήρξε θέμα προθεσμίας κατάθεσης ε, προτάσεων για τροποποιήσεις ή αλλαγές υπευλήθησαν με καθυστέρηση και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από πλευρά τη λέγει ότι έκανε ό,τι έπρεπε, έκανε όλα όσα έπρεπε να είχε πράξει και ότι ε, είχαν όλα παρασχεθεί έγκαιρα. Αν τώρα ε, δεν θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει δίκιο η επιχείρηση, το δικαστήριο δεν συμμερίστηκε τις απόψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεώρησε όμως ότι είχε βλαφθεί η εταιρεία και η εταιρεία που ζητούσε αποζημίωση έπρεπε να ε, της καταβληθεί. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι η αντιστάθμιση, μια και το ποσό περιορίστηκε, δεν ήταν η αρχικά προβλεπόμενη αντιστάθμιση, όμως πρόκειται για ένα αρκετά μεγάλο κονδύλιο πιστεύω εγώ έτσι λοιπόν τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το θέμα θεωρεί ότι εκκρεμεί ακόμη, μια και βρίσκεται υπό ε, εξέλιξη η άσκηση προσφυγής, έχουν εφεσιβάλει και θα ληφθεί απόφαση επ' αυτής της προσφυγής στο μέλλον από πλευράς του δικαστηρίου. Λέγει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το δικαστήριο θα μπορούσε ίσως να συμφωνήσει με τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς δεν μπορούμε να προδικάσουμε, πρέπει να αναμείνουμε και να δούμε τι θα γίνει. Συνιστούμε υπέρ της μεταφοράς των κονδυλίων αυτών Λυπούμε για την κατάσταση που διαμορφώθηκε με τον τρόπο που διαμορφώθηκε, όμως από όσα γνωρίζουμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και έχουμε συναγάγει και από τα έγγραφα, φαίνεται ότι αμφότερες οι πλευρές είχαν θετικά επιχειρήματα για να θεωρούν ότι η δική τους στάση και συμπεριφορά ήταν η ορθή. Όμως σε αυτή τη χρονική στιγμή αυτό αποβαίνει εις βάρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια και η απόφαση ήταν εις βάρος της. Συζήτησα ένα θέμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνέπησαν ότι άλλαξαν οι όροι και οι προϋποθέσεις σε σχέση με τις συμβάσεις. Μια νέα σύμβαση που έχει συναρθεί με ε, διάφορους ε, ενδιαφερόμενους, αυτό όμως δεν μπορεί να υπάρξει αναδρομικά, δεν είναι δυνατόν κάποια αλλαγή να ληφθεί υπόψη αναδρομικά, όμως οι νέες συμβάσεις, τα νέα συμβόλαια είναι διαφορετικά εφ' Γι' αυτό είμαι υπέρ αυτής της μεταφοράς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Πόρτας παρακαλώ. Μόνο και μόνο ήθελα μία ερώτηση να διατυπώσω αν γίνεται. Γιατί δεν κατάλαβα απόλυτα καλά. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα ζητά να ασκηθεί προσφυγή, έχει εφεσιβάλει, ή γιατί πρέπει να πληρώσει τώρα, να καταβάλει αυτά τα ποσά τώρα. Αυτή είναι ερώτησή μου, αν μπορείτε να την απαντήσετε παρακαλώ. Euh, on demande Θέλετε εσείς να απαντήσετε, ε, Συντόνια, η, η Κομισιόν. Προσέξτε, έλεγξα και εγώ το εξέτασα αυτό γιατί και εμένα με ενδιέφερε το θέμα αυτό. Η απόφαση, η νομολογία του δικαστηρίου ποια ήταν είναι non-suspensive, δεν άρει, δεν μπορεί να άρει στα γαλλικά. Δηλαδή πρέπει να πληρωθεί, να καταβληθεί αυτό το ποσό πριν από την άσκηση προσφυγής και εφόσον δεν θα έχει ακόμα τοποθετηθεί επί της προσφυγής ε, το δικαστήριο, αν τοποθετηθεί αντίθετα θα πρέπει να επιστραφούν αυτά τα κονδύλια. Και πού. Ζούμε λοιπόν αυτή τη μεταφορά υπέρ, κατά δεν έχουμε εποχές. Επομένως αυτή η μεταφορά πιστώσεως εγκρίνεται. Τώρα, άλλες μεταφορές πιστώσεων που αφορούν, ε, που την, την εισηγήτρια. Σας λέμε για ενημέρωσή ότι θα πάμε για 15 Μαρτίου και όχι σήμερα. Επομένως τώρα συνεχίζουμε για στις άλλες μεταφορές πιστώσεων που αφορούν την Χέλγα. Συζητήσαμε προ λίγο για αυτή τη μεταφορά πίστωσης για την εξωτερική υπηρεσία και επομένως θα προχωρήσουμε για τις άλλες. Χέλγα. Για τις άλλες μεταφορές, Χέλγα. Ευχαριστώ. Ξεκινώ με το ελεγκτικό συνέδριο, λοιπόν. Ο Γενικός Γραμματέας του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκανε μια συνολική ε, εξέταση πώς παρέχεται η υπηρεσία σε σχέση με την ασφάλεια και σε σχέση με το θεσμικό μας όργανο. Κατέληξε στο ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι για την ασφάλεια είναι με υπηρεσίες in-house resources. Έτσι καταργήθηκε η σύμβαση με τον πάροχο υπηρεσιών και στελεχώνεται με ένα μικρό αριθμό παρόχων αντι, αντιμετωπίζοντας τους στόχους για την ασφάλεια αυτό θα οδηγήσει λέμε ε, σε εξοικονόμηση πάνω από 100.000 ετήσια. Οι υπηρεσίε για την ασφάλεια πληρώνονται από το κονδύλιο 2026 ασφάλεια εποπτεία κτηρίων. Από το Μάρτιο 2011 ένα σημαντικό κονδύλιο θα επιμερίζεται στο 1400 κονδύλιο και για τα στελέχη ιδιαίτερα υπό το 1406 συμβατικά εργαζόμενοι. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να μεταφερθεί το ποσό που ζητείτε. 320.000 ευρώ λοιπόν από το 2026 στο 1400 κονδύλιο, υπαριθμό 1400. Συνιστώ λοιπόν να είμαστε υπέρ αυτής της μεταφοράς. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Δεν ζητά κανείς το λόγο. Υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται μεταφορά. Επόμενη μεταφορά, Χέλγα. Επόμενη μεταφορά, Χέλγα. Ναι, είναι το πρόγραμμα για τον διαμεσολαβητή ζητεί μεταφορά μιας προσωρινής α5 ε, θέσεως εργασίας σε μόνιμη θέση εργασίας. Επιχειρηματολογεί και λέει ότι αυτό θα οδηγήσει στο να αποφύγουμε ευμεταβλητότητα όσον αφορά νομομαθείς γλωσσομαθείς ε, μεταφραστές. Είναι δύσκολο με ένα τέτοιο προφίλ να διατηρηθούν στελέχη με προσωρινή σύμβαση εργασίας. Είχα μια ευκαιρία πέρσι να συζητήσω με τους αρμόδιους υπεύθυνους και είναι δικαιολογημένο το αίτημα και συνιστώ να εγκρίνουμε υπέρ τη μεταφορά κονδυλίου και να υπερψηφίσουμε. Αλλαγή κατηγορία. Ποιο είναι υπέρ αυτή τη μεταφορά. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Χέλγα. Next. Χέλγα, επόμενη μεταφορά, έτοιμα μεταφοράς. Κοινοβούλιο, C1, 30 θέσεις θα απελευθερωθούν από το αποθεματικό. Ο στόχος αυτού του εγχειρήματο είναι να ζητηθεί η απελευθέρωση 726.000 ε, ευρώ όσον αφορά τον τίτλο 1 άτομα που εργάζονται σε αυτό το θεσμικό όργανο από το κεφάλαιο 100 προσωρινά, προσωρινές ε, πληρωμές αφορά 30 στελέχη 740.026 ευρώ που είχαν ζητηθεί από το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους. Ζήτησε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση αυτού του κονδυλίου το Κοινοβούλιο. Οι αντίστοιχες πληροφορίες δόθηκαν, αλλά πολύ πρόσφατα μόνο. δυστυχώς. Και γι' αυτό θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε κάπως περισσότερο χρόνο. Πρέπει να αναβάλουμε την πληροφορία, διότι αυτά τα στοιχεία υπευλήθησαν με μεγάλη καθυστέρηση, πολύ πρόσφατα. Καλό θα ήταν να αναβάλουμε την ψηφοφορία, να αποφασίσουμε υστερότερα. Είμαι στις διαταγές σας, ε, κύριε Συγκεφρή. Αν δεν έχετε αρκετέ πληροφορίε, θα κάνουμε ό,τι κάναμε και προηγουμένω για το σπίτι τη ευρωπαϊκή ιστορία. Αναβάλουμε την ψηφοφορία, προλαβαίνουμε. Ούτω ή άλλω. για το C3 η Helga Trooper λοιπόν το, ε, η επιδότηση για βοηθούς πρόταση είναι να ζητηθεί η απελευθέρωση 30 εκατομμυρίων χιλιάδων όσον αφορά τις πληρωμές για το 420 για τους βοηθούς από το κεφάλαιο 100 προσωρινές πληρωμές όσον αφορά την κατάθεση των αναγκαίων πληροφοριών που δόθηκαν όσον αφορά το επίδομα βοηθών είναι το δεύτερο, η δεύτερη δόση της αύξησης ε, του επιδόματος βοηθών που αφορά τα 1.500 ευρώ αναμέλος αναμήνα για τους ευρωβουλευτές. Θα ήθελα επ' αυτού να πω τα εξή. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε λόγο για αυτό το θέμα που είναι αρκετά περίπλοκο ως θέμα. Γνωρίζετε ότι εγώ είχα επιχειρηματολογήσει για την πρώτη, το πρώτο αίτημα συνδρομής και είχα πει λόγω Λισαβόνας έχουμε νέες αρμοδιότητες, νέο φόρτο εργασίας, πρέπει να ανταποκριθούμε. Τώρα όμως θα ήθελα να πω ότι όπως γνωρίζετε πάντα ήμουν διστακτική και δεν ήμουν υπέρ της δεύτερης δόσης, υπέρ καταβολής δεύτερης δόσης. Τώρα έχουμε κάποια στοιχεία που λένε ότι μόνο 70 νέες τέτοιες θέσεις βοηθών στελεχώθηκαν. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ διστακτικοί και πάλι αν πραγματικά χρειάζεται αυτή η επιδότηση ουσιαστικά. Επανέρχομαι στη συζήτηση που είχαμε και προηγούμενα μόλι για τον Ευρωπαϊκό Οίκο Για να είμαι ξεκάθαρη και ειλικρινή. Αν υπάρχουν τόσοι πολλοί λόγοι να είμαστε υπέρ τη δημιουργία τη προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Οίκου από την άλλη φορά, αν θέλουμε να πούμε ότι είμαστε πρόθυμοι για εξοικονόμηση κονδυλίων, υπό το δικό μου πρίσμα προσωπικά, είναι η δική μου άποψη, αλλά είναι και η άποψη τη πλειοψηφία των μελών, θα μπορούσε να υπάρξει ένα συνδυασμό και των εξοικονομήσεων και των ε, προτεραιοτήτων μας για να πούμε θα έχουμε προτεραιότητα τον Ευρωπαϊκό Οίκο Ιστορίας ή πρέπει να βρεθούν και άλλες περικοπές ή εξοικονομήσεις κονδυλίων τουλάχιστον προς όφελος της μελλοντικής συζήτησης που θα γίνει κατά τα τέλη Μαρτίου. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για παγίωση σε υγιή βάθρα του προϋπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του Επιτρόπου Λεβαντόφσκι πρέπει να βρούμε μια πολύ καλή ισορροπία για τα θέματα των κονδυλίων του προϋπολογισμού. Γι' αυτό θα έλεγα δεν είναι η καλύτερη χρονική συγκυρία να το κάνουμε σήμερα και να εγκρίνουμε αυτή την επιδότηση για βοηθούς. Να τα συνδυάσουμε με τη γενικότερη εικόνα στο μέλλον. Σύστασή μου να αναβάλουμε την ψηφοφορία και να επανέλθουμε υστερότερα. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ μου ζήτησαν το λόγο. Η Χέλγα προτείνει να αναβάλουμε τη συζήτηση, την απόφαση μάλλον. Οπότε ίσως μπορούμε να αναβάλουμε και τη συζήτηση, διότι δεν θα έχουμε χρόνο και για τα υπόλοιπα. Δεν μπορούμε λοιπόν να αναβάλουμε, οπότε θα δώσω το λόγο σε όσους τον ζήτησαν. Γκόραν, όπως γνωρίζετε όλοι αυτό το θέμα είναι κάτι εξωγήν επίμαχο. Ο κύριος Άλβαρο το έθεσε όταν έκανε την ε, δήλωση σχετικά με την ψηφοφορία προηγουμένως και εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτό το επίδομα για τους συνεργάτες δεν είναι μόνο για απασχόλησή τους ή στις Βρυξέλλες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την βελτίωση της θεσεώς τους για πρόσληψη αλλού συνεργατών. Αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο γιατί υπάρχει μια σχέση στενή μεταξύ αυτού του, του, του, του κονδυλίου και των κονδυλίων για τα νέα κτίρια. Εμείς είμεθα υπέρ ως πολιτική ομάδα αυτών των ε, αυτών των κονδύλιων. Για αυτά τα 1500 και θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι το να δώσουμε εδώ το πράσινο φως δεν προδικάζει το τι θα πούμε για το νέο κτίριο όπου επιφυλασσόμεθα ακόμη. Οι περισσότεροι στην πολιτική μας ομάδα πάντως είναι υπέρ της εκταμείευσης αυτού του ποσού. Και επομένως θέλετε να ψήσουμε τώρα. Ναι, ναι, ναι, λέει κύριε Χάουκ. Πόρτος. Θα ήμουν υπέρ τη αναβολή ψηφοφορία και αναβολή τη συζήτηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάτι τέτοιο. Όλη αυτή η συζήτηση λοιπόν για τα χρήματα, για τα κονδύλια αυτά, για τους βοηθούς των Ευρωβουλευτών. Από την αρχή είχε πάρει στραβή πορεία και εξέλιξη ξεκινώντας με τα 1.500 ευρώ ετήσια και 1.500 τον επόμενο ε, χρόνο και τα αποτελέσματα για την επίτευξη των στόχων δεν δικαιολογούνται από κάτι τέτοιο. Με 1.500 ευρώ δεν μπορεί να προσλάβει κανείς άτομα τα οποία να είναι κατάλληλα ως βοηθή. Αλλά κυρίως δεν μπορώ να κατανοήσω, δεν καταφέρνω να κατανοήσω καθόλου πώς είναι δυνατόν η πλειοψηφία των συναδέλφων που έχουν θέσει τόσο στεναρέ και αποφασιστικέ υπέρ πολιτικών αυστηρότητα και πειθαρχία να αυξάνουν και να δείχνουν κατανόηση για πολιτικέ αύξηση. Όταν έχουμε πολιτική περικοπών και αυστηρότητα δημοσιονομική, εξ ονόματο του ευρωπαϊκού επίπεδου, ευρωπαϊκού Προπολογισμού και στα εθνικά ε, κοινοβούλια, Πώ είναι δυνατόν για τη διάθεση τέτοιων κονδυλίων να έχουν διαφορετική άποψη. Αλλάζουν άποψη, τι γίνεται δεν μπορώ να το κατανοήσω αυτό. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και κάθετοι επ' αυτού. Ε, Δεν ξέρω αν υπάρχει ισοδυναμία στις υπόλοιπες γλώσσες, αλλά στους Γάλλους καθολικούς λέμε ότι για να είναι κανείς ελεήμων πρέπει να ξεκινά από τον εαυτό του. Και στην Πορτογαλία έχουμε μια έκφραση που λέει ότι όποιος μοιράζει και τα δίνει και δεν παίρνει το καλύτερο κομμάτι για τον εαυτό του εντάξει να μην δώσουμε συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση κύριε Φερνάντες Παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο δεν ακούγεται eh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα αυτά τα κονδύλια για τα οποία κάνουμε λόγο δεν είναι για εκείνον που τα μοιράζει και τα ξαναμοιράζει. Αυτά για τα οποία κάνουμε λόγο είναι για τους βοηθούς, εντάξει, και όχι για ίδιο όφελο και για την επίτευξη των στόχων που καθορίσαμε βελτίωση στην νομοθετική εργασία μας. Αλλά επίσης είναι ένας, μια δέσμευση που είχαμε αποφασίσει. Είπαμε 3.000 ευρώ αύξηση. θα έχουμε σε δύο φάσεις για να μην υπερβαρυνθεί ο προϋπολογισμός. Η πρώτη δόση αποφασίστηκε, εγκρίθηκε 1.500 ευρώ. Η δεύτερη δόση είναι συμβιβασμό. Δεν έχει νόημα να κάνουμε μισό συμβιβασμό, να πούμε ε, τα 1.500 ευρώ να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2011 αναμένοντας λέει πληροφορίες, πληροφορίες σαφείς, πληροφορίες που θα ανταποκρίνονται σε αυτό το οποίο είχαμε εμείς ε, ζητήσει. Και γι' αυτό είναι αυτό μια συζήτηση που έχει γίνει ήδη πολλές φορές στο παρελθόν. Και μπορούμε χωρίς κανένα πρόβλημα να αποφασίσουμε, να εγκρίνουμε τη μεταφορά αυτό, αυτή για ένα θέμα που δεν είναι καινούριο και που είναι ανταπόκριση σε υποχρεώσεις που είχαμε αναλάβει. Ευχαριστώ κύριο Σάγκλον. Yes, Chairman, just briefly. Uh, Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Η δική μας ομάδα συστηματικά είναι κατά δεύτερη ε, μεταφοράς για, τη, για τους βοηθούς. Εδώ θα στηρίξουμε λοιπόν τον συγκεκριτή στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ε, νεαρά Ίγκια Γκρέσλερ μπορεί κανείς να επιστήσει την προσοχή αν θέλετε ότι για αυτές τις δαπάνες έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία να μην τα δαπανίσουμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δαπανίσουμε αυτά τα κονδύλια. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν πάρα πολλή δουλειά και πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν, να εργάζονται όπως πρέπει, με αξιοπρέπεια. Όλοι αξίζουν αυτή τη δαπάνη εφόσον έχουν ανάγκη. Αλλά δεν δέχομαι την υποκρισία ο να αφήνουμε πράγματα να εξελίσσονται όποια και να είναι και όταν έρχεται η ώρα του λαϊκισμού να λέμε όχι, αυτέ οι δαπάνε δεν θα γίνουν. Την πολιτική δουλειά που πρέπει να κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να την κάνουμε αν δεν έχουμε περισσότερου βοηθού. Εγώ ίδια στο γραφείο μου, γιατί κάθε έκθεση πρέπει να τη συντάσω αλλιώ η ίδια, ή αγγλικά ή γαλλικά. Και γι' αυτό θέλω να, να επισημάνω ότι κάποιο που δεν χρειάζεται τέτοια βοήθεια, δεν χρειάζεται αυτό το κονδύλιο. Έχω αυτά τα καλά μαντάτα. Μπορεί κανεί να τα δώσει αυτά τα κονδύλια για τη δίκηση του Κοινοβουλίου για τα κτίρια στο Λουξεμβούργο ή αλλού, στο mopping up, δηλαδή στα γάλ, στα υπόλοιπα υποκαθάριση μπορούν να συναθρίζονται αν δεν τα χρειάζονται οι ευρωβουλευτέ. Να μην μακρύνουμε αυτή τη συζήτηση. Αυτό είναι όμω μέρο αυτή τη αλήθεια που πρέπει να δούμε. Και για τα άλλα θεσμικά όργανα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο, όταν επιτρέπουμε πράγματα να γίνονται που ποτέ δεν θα επιτρέπαμε στον εαυτό μα, ε, τότε πώ θα είμαστε δημοσιονομικοί ελεγκτέ που θα αξίζουν το, ε, ε, τα λεφτά τους. Πού θα είμαστε όταν θα πρέπει κάπου να ελέγξουμε στις εξωτερικές δράσεις, σε άλλες δαπάνες, για πολιετής δαπάνες και μεγάλα κονδύλια που θα πρέπει να περικόπτονται. Πότε θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι των λόγων που δίνουμε όταν ελαφρά την καρδία δαπανούμε εκατομμύρια ή δεσμεύουμε εκατομμύρια για μεγάλο χρονικό διάστημα επί πολλά έτη. Δεν είναι δυνατόν από τη μία πλευρά να κάνουμε κάτι για μεγαλο χρονικο διαστημα επι πολλα ετη δεν ειναι δυνατον απο τη μια πλευρα κανουμε κατι τετοιο και να μην δίνουμε από την άλλη πλευρά τα χρήματα για τους βοηθούς. Να αφαιρέσουμε τη δυνατότητα να δουλεύουμε καλά δεν είναι δίκαιο. Ας κάνουμε αυτό που χρειαζόμαστε. Να δώσουμε τα κονδύλια να δουλεύουμε σωστά. Αλλιώς δεν μπορούμε να είμαστε σωστοί ευρωβουλευτές όπως αναμένουν οι πολίτες από μας Ευχαριστώ. Είναι σαφής η τοποθέτηση να μην ξαναρχίσουμε όλη τη συζήτηση. Τελευταίος ο κύριος Γκάιερ, παρακαλώ. Λοιπόν, επί της ουσίας Όλα αναφέρθηκαν. Έτσι, όσα είναι υπέρ της έγκρισης, της απόφασης κτλ. Δύο συζητήσεις θέλω να αναφέρω, δύο στοιχεία. Πρώτο σημείο σε μία από τις πρώτες ψηφοφορίες που συμμετείχα σε αυτή την κοινοβουλευτική επιτροπή ήταν η αγορά του ΤΕΦ1. Αν θυμάμαι καλά, αυτό επιχειρηματολογήθηκε με τον τρίτο λέει βοηθό στις Βρυξέλλες. Ναι, σε πόσα άλλα γραφεία θα έχουμε όμως βοηθούς που θα καταλαμβάνουν αυτά τα γραφεία. Το αναφέρω εδώ. Μπορεί κανείς να ενοικιάζει χώρους όταν δημιουργηθεί μία νέα, αν θέλετε, διασύνδεση μεταξύ οίκου ιστορίας και επιδόματος ε, για τους βοηθούς, τότε είμαι υπέρ της επικέντρωσης στις κυριότερες ευθύνες μας. Τότε οι κυριότερες ευθύνες μας είναι να νομοθετούμε και τι, να ανοίγουμε και μουσεία. Παρακαλώ οι συνάδελφοι να είναι κάπως περισσότερο ειλικρινείς και λίγο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να έχουν. Διότι εμείς εκπροσωπούμε 550 εκατομμύρια πολιτών νομοθετικά με το έργο μας ως αιρετοί εκπρόσωποι των πολιτών έναντι του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να μου πει κάποιο πώ με αυτά τα 1500 ευρώ τα οποία θα απελευθερωθούν τώρα θα προσλάβω τον τρίτο βοηθό. Είναι απόλυτα σωστό αυτό το οποίο είπε ο Γιώραν Φάρμ. Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο με αυτό, να διαθέσουμε ε, διαφορετικά αυτά τα κονδύλια. Να πάρουμε μη ακαδημαϊκούς, μη πανεπιστημιακούς αποφύτους. Εντάξει, αν κάποιο θέλει όμως σε αυτό το σώμα στο Ευρωκοινοβούλιο να γίνεται σωστή νομοθετική δουλειά, δεν μπορεί να διασφαλιστεί αυτή η, νομική, η νομοθετική δουλειά αν εμεί περικόψουμε τι δυνατότητε να είμαστε σωστοί ευρωβουλευτέ με του αναγκαίου βοηθού. Ευχαριστώ. Συμπεραίνω από όλη αυτή τη συζήτηση ότι η πλειοψηφία των ε, συναδέλφων θέλουν να ψηφίσουμε τώρα με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΥΤΗ. Ε, μάλλον με τη μη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΥΤΗ. Εδώ λοιπόν θα ψηφίσουμε για αυτήν την ε, μεταφορά, την απελευθέρωση πιστώσεων τέλο πάντων. Ε, υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Δεν υπάρχουν αποχές. Σαφή ψηφοφορία. Είχαμε και τι εξηγήσει. Η απόφαση ελήφθη. Ε, Δεν έχουμε παρά μόνο λίγα λεπτά και έχουμε πολλά θέματα ακόμη. Στρέφουμε προς την Μόνικα. Μόνικα, Πρέπει να το θέσετε τώρα το θέμα ή μπορείτε να το, να το πείτε και την επόμενη φορά. Το σημείο 20. Σοφία, θέλετε να το σχολιάσετε τώρα ή μπορούμε να το αναβάλουμε για την επόμενη. Το αναβάλουμε. Ωραία. Όχι, δεν μπορείτε. Τότε δύο προτάσεις μόνο. Ich kann maximal bis 15, aber es geht auch innerhalb von zwei σε δύο λεπτά μπορώ επί της ουσίας να τοποθετηθώ. Σε δύο λεπτά μπορεί να γίνει. Διότι γνωρίζουμε το χαρτοφυλάκιο από πέρυσι ήδη. Και μάλιστα πρόκειται για το Γραφείο Πληροφοριών στη Σόφια. Πολύ γοργά μπορούμε να το κάνουμε έχουμε τα πιο απίθανα κτίρια που δεν μπορούν να είναι προσπελάσιμα για τους πολίτες. Γι' αυτό τον λόγο θα αγοραστεί ένα νέο κτίριο. Εποφελούμαστε εμείς από αυτό. Μια και η αγορά κινήτων στη Βουλγαρία έχει μειωμένες τιμές και σε μεγάλο ε, ποσοστό κιόλα λόγω της οικονομικής κρίσης. Έτσι λοιπόν το κόστος το οποίο προβλεπόταν στα 13 εκατομμύρια για την αγορά ενός τέτοιου κτιρίου θα είναι 9 εκατομμύρια τώρα με το opting out και opting in. Και έτσι θα έχουμε ένα επαρκές επίπεδο επίπεδο εμβαδού και χώρων στάθμευση. 60% θα επιστρέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του συνολικού κόστου και τα έχουμε συζητήσει αυτά πέρσι. Παρακαλώ να εγκριθεί αυτό γιατί τα κονδύλια αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα μέχρι τέλη Μαρτίου. Ολοκλήρωσα. Ευχαριστώ. Η συγκήτριά σας λοιπόν λέει να συμφωνήσουμε, το εγκρίνουμε. Δεν υπάρχουν διαφωνίες. Ακολουθούμε λοιπόν την άποψη της συγκήτριας. Τώρα μας μένουν δύο θέματα. Μπάρμπαρα πρώτα απ' όλα, σε χαιρετώ. Θα της δώσουμε πέντε λεπτά για να, τις, για να παρουσιάσει τα σημεία 7 και 8. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης ε, για την Τσεχία και την Πολωνία. Μπάρμπαρα, ευχαριστώ πρόεδρε. Σήμερα με μεγάλη μου χαρά σας παρουσιάζω την κινητοποίηση του Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσαρμογής για την παγκοσμιοποίηση για τα δύο πρώτα χρόνια. Εδώ για το 2011 έχουμε κινητοποίησει για δύο κράτη, την Δημοκρατία της Τσεχίας, συγκεκριμένα για τους απολυμμένους της πολυεθνικής Unilever και την Πολωνία σε ό,τι αφορά την, περιοχή, την ε, επαρχία του Πόντ Καρπάκη. Ε, ελπίζω να το προφέρω σωστά. Σε ό,τι αφορά την ε, αίτηση της Τσεχίας, αφορά τους 634 εργαζομένους που απασχολούνταν στο λιανεμπόριο στην, και στην βιομηχανία στην επαρχία του Στρέτζιντσέκη. Μιλάμε για 30 εκατομμύρια ευρώ εδώ, ενώ σε ό,τι αφορά την Πολωνία οι απολύσει φτάνουν τις, ε, τους 594 εργαζομένους από τρεις εταιρείες στον τομέα των, ε, της κατασκευής μηχανημάτων. Το ποσό, ποσό που ζητάτε είναι 453 εκατομμύρια ευρώ. Συγγνώμη, 453.000 ε, ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πω ότι εδώ έχει ζητήσει μοίρια ε, ευρώ για την δημοσιονομική γραμμή που απευθύνονται σε αυτό το ταμείο. Οπότε εδώ χαιρετίζω την, την, την ε, πίστη που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το Ταμείο. Εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο όλοι θα κινητοποιηθούμε για το μέλλον του Ταμείου και θα δούμε τι σημασία θα λάβει τα επόμενα χρόνια. Θα δούμε εάν στο άμεσο μέλλον θα μπορέσουμε να διοργανώσουμε συζήτηση και σε αυτή την Επιτροπή, διότι εδώ ήθελα να σας επισημάνω ε, ξανά και να δώσω έμφαση στο πόσο σημαντικό είναι το Ταμείο αυτό. Ε. Τέλεια. Θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε ξανά επί της ουσίας για τον επιπλέον λόγο ότι οπωσδήποτε από την πλευρά του Συμβουλίου θα συναντήσουμε υπουργού. Υπουργού για να κινητοποιηθεί το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και οι κατεπήγουσες βοήθειε με επιστώσεις πληρωμών και δυσκολίες ανάλογες με αυτές που είχαμε διαπιστώσει για το Ταμείο Αλληλεγγύη. Ξέχασα να σα πω ότι η ψηφοφορία για τα θέματα αυτά στην Επιτροπή Προπολογισμού θα γίνει στι 16 Μαρτίου, ενώ στην Ολομέλεια η έγκριση προβλέπεται τον Απρίλιο. Δεν ξέρω την ημερομηνία για την ε, υποβολή τροπολογιών. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν. Ελπίζω όμω, και εφόσον υπάρχουν θα είναι καλοδεχούμενες. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών έχει οριστεί για τις 4 Μαρτίου αύριο στις 10. Δεν θα είναι πολλές προφανώς. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε την Μπάρμπαρα. Οπότε περνάμε στο τελευταίο σημείο. Πρόγραμμα στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Ο Ντομινίκ Ρικέ που βλέπει τη θάλασσα από τη Βαλανσιέν ε, πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομο, αφού είμαι και τελευταίο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τι προπαρασκευαστικέ δράσει και το πιλωτικό σχέδιο που ολοκληρώθηκαν το 2010, προκειμένου η θαλάσσια πολιτική να ε, οριστεί στο δημοσιονομικό πλαίσιο του 2011 στο 2013 με 50 εκατομμύρια ευρώ. Η συγκεκριμένη έκθεση αφορά τους στόχους του προγράμματος και με κεντρική ιδέα ότι οι στόχοι αυτοί πρέπει να τύχουν ε, πιο συγκεκριμένη διευθέτηση ω προ τι δαπάνε. Και να συμμετάσχει στην εκτέλεση και τον έλεγχο τη εκτέλεση το Κοινοβούλιο. Κυρία Γκρολιέ, έχει υποβάλει τροπολογίε για το κείμενο. Μπορέσαμε μαζί να συνεργαστούμε αποτελεσματικά. Προτείνω λοιπόν να αποδεχτούμε τις τροπολογίε αυτές έχουμε ετοιμάσει για τι τροπολογίε 4, 10 και 11 συμβαστική τροπολογία. Είναι σημαντικό λοιπόν νομίζω στο κείμενο αυτό να διευκρινιστεί ποιε είναι οι δύο δημοσιονομικέ γραμμές που ορίζονται. Εδώ προσδιορίζουμε ότι στο ενδιάμεσο θέλουμε να κάνουμε μια αποτίμηση του αντικτύπου και με τροπολογίε να μπορούμε να διορθώσουμε τον προπολογισμό για τη χρηματοδότηση αυτή τη νέα πολιτική. Την οποία προτείνουμε βεβαίω να στηρίξουμε. Εδώ να θυμίσω ότι για τι δημοσιονομικέ πτυχέ τοποθετείται η Επιτροπή μα, ενώ για τα θέματα επί τη ουσία τοποθετείται η Επιτροπή, Μεταφορών. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, αλλά καθότι είστε αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών, είστε στην κατάλληλη θέση για να φροντίσετε ώστε η δική μα απόφαση τη 15 η 16 μαρτιου να ληφθεί απόψη από την Επιτροπή Μεταφορών. Τι χαρά σα θέλετε να εκφράσετε. Ε, ναι, Πρόεδρε, γιατί όχι. Ε, μπορέσαμε να συνεργαστούμε πολύ καλά με τον κύριο Ρίκε. Ε, ίσως βλέπω περισσότερο τη θάλασσα από ότι εκείνο, ε, από την Αμιά, από ότι από τη Βαλανσιέν. Και νομίζω ότι συνεργαστήκαμε τόσο καλά. Το κείμενο είναι πραγματικά ισόρροπο και εκφράζει την επιθυμία μα να δούμε την πολιτική αυτή να προκοδοτείται με έναν επαρκή προπολογισμό. Ίσως όταν μένει κανείς σε περιοχές ε, της ε, ξηράς ε, που δεν είναι κοντά στη θάλασσα, δεν τα αντιλαμβάνεται αυτό τόσο καλά, αλλά είναι σημαντικό να είναι πλήρης ο προπολογισμός της θαλάσσιας πολιτικής. Ναι, και εγώ, εφόσον προέρχομαι από παράκτια όλοι, έχω ιδιαίτερη εκτίμηση για το θέμα αυτό. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι είναι συνενετική η προσέγγισή σας, πολύ καλό αυτό. Δεν υπάρχουν άλλε τοποθετήσει. Θα το ψηφίσουμε στην επόμενη συνεδρίασή μα. Σα ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Είχαμε μια πολύ φορτωμένη σε διάταξη, αλλά καταφέραμε να τελειώσουμε και 10 λεπτά νωρίτερα. Σα δίνω ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο για την Ολομέλεια. Και για την ερχόμενη συνεδρίασή μα στι 15 Μαρτίου. τη συνεδρίαση.